Uh, we to start the meeting because time Να μην χάνουμε λοιπόν το χρόνο μας που είναι πολύτιμος και επομένως να ξεκινήσουμε αμέσως με την ε, ε, ακρόασή μας όσον αφορά την νομοθετική δέσμη μέτρων. Θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα ε, με δύο εκπροσώπους ε, μελετητές ε, εμπειρογνώμονες. Θα ακούσουμε πρώτα τον καθηγητή κύριο Μπάχτλερ και τον κύριο Κάρλος Μέντες από το, Ευρωπαϊ... από το Ερευνητικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Πολιτικών, EPRC. Θα ακούσουμε λοιπόν αυτούς τους δύο συναδέλφους και μετά θα δούμε, θα ακούσουμε μάλλον τον επικεφαλής ε, οικονομολόγο του ε, Κέντρου Ευρωπαϊκής Πολιτικής, τον κύριο Ζούλεγκ. Θα εστιαστούμε λοιπόν πρώτα σε αυτές τις δύο παρουσιάσεις και μετά θα προχωρήσουμε ε, στις παρουσιάσεις των άλλων εμπειρογνωμόνων. Τζον, Τζον Μπάχτλερ μαζί με τον ε, Κάρλος Μέντες αν μπορείτε να ξεκινήσετε λοιπόν και να μας ε, υποβάλλετε ε, τα συμπεράσματά σας σχετικά με, την, με τις επιλογές που θα έχουμε όσον αφορά την πολιτική συνοχής. Μακάρι να είχαμε ώρες ολόκληρες να σας ακούσουμε, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε παρά 20 λεπτά, 15 λεπτά μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι σίγουρη ότι μετά από τα 15 λεπτά θα μας ευγνωμονείτε που είχαμε μόνο 15 λεπτά χρόνο στη διάθεσή μας. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε και με χαρά μας θα συνεισφέρομαι σε αυτήν την ε, ε, ε, συνάντηση. Και ο, εγώ ίδιος και ο συνάδελφος Κάρλος Μέντες εκπροσωπούμε το EPRC και δουλεύουμε ε, για τα θέματα αυτά εδώ και καιρό. Έχουμε, ε, μας έχει ανατηθεί να μελετήσουμε την ε, αναθεωρητική νομοθετική δέσμη μέτρων στα πλαίσια της πολιτικής για τη συνοχή. Εγώ θα ήθελα σήμερα κυρίως να επικεντρωθώ στα ζητήματα αυτά τα οποία ε, αφορούν την στρατηγική συνοχή καθώς επίσης και θέματα που αφορούν την αποτελεσματικότητα και την ε, απλούστευση των διαδικασιών γιατί θεωρούμε ότι αυτά είναι ε, ένα από τα κύρια στοιχεία τα οποία θα μας οδηγήσουν σε αυτήν την διαδρομή. Έχουμε και κάποιες διαφάνειες τις οποίες νομίζω ότι έχετε και εσείς στη διάθεσή σας και βεβαίως οι συνάδελφοι θα δουν ε, και τις διαφάνειες στην ε, οθόνη. Μέχρι όμως να λειτουργήσει η οθόνη θα ήθελα να σας πω το εξής. Κύριος στόχος της ε, έρευνας αυτής ήταν η αξιολόγηση του πακέτου που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς επίσης και κάποια μέτρα που αφορούν τον προϋπολογισμό ε, χωρίζεται σε έξι ε, κατηγορίες, έξι κεφάλαια που ασχολούνται με τελείως διαφορετικά θέματα το ένα με το άλλο, δηλαδή ε, την διάσταση του χώρου, την στρατηγική, την στρατηγική συνοχή και τον προγραμματισμό, την απόδοση, την επίδοση, την διασφάλιση και την απλούστευση κτλ. Ε, και ε, ε, επ' αυτών θα κάνουμε και κάποιες προτάσεις και συστάσεις και προς το Κοινοβούλιο ξεκινώντας με την αρχιτεκτονική. Υπάρχει μια διαφάνεια που δεν τη βλέπω ακόμα. Είναι λίγο πιο μετά από αυτή που δείχνετε τώρα. Η κατάθμιση των πόρων για την επόμενη προγραμματική περίοδο ε, σε σύγκριση και με την προηγούμενη περίοδο 2007-2013. Φαντάζομαι ότι είναι στοιχεία τα οποία σας είναι ε, οικεία, δεν υπάρχουν πάρα πολλοί και, και εκεί είναι οι μεγάλες ε, αλλαγές. Όσον αφορά αυτήν την οικονομική κατάτμιση πρέπει να σας πω ότι στην μελέτη μας κάναμε μια αναλυτική χαρτογράφηση και των επιπτώσεων της πρότασης και όσον αφορά την κατανομή των ε, πόρων αλλά και όσον αφορά την επιλεξιμότητα. Ε, βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει αστάθεια όσον αφορά τα στοιχεία. Μέχρι τώρα βασίσαμε τους προϋπολογισμούς μας στα στατιστικά στοιχεία του 2011 ε, που έδιναν ε, στοιχεία ΕΠ για το 2006-2008 αλλά είχαμε ε, πλέον και καινούρια στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν σημαντικές διαφορές γιατί περιλαμβάνουν ε, στοιχεία ΑΕΠ και για το 2009. Βλέπουμε λοιπόν σε αυτά τα νέα στοιχεία σημαντικές διαφορές όσον αφορά την επιλεξιμότητα. Ας πούμε εκτιμούμε ότι ακόμα έξι περιοχές επιλέξιμες για λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, τρεις εκ των οποίων ε, στην Ελλάδα. Υπάρχουν 8 περιοχές πλέον ως μεταβατικές περιοχές για το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα και την Ισπανία που ήταν παλιά πιο ε, ανεπτυγμένες, δηλαδή επιλέξιμες για, ε, για, για, για καθεστώς πιο ανεπτυγμένες περιοχής. Επίσης, δύο περιοχές πλέον γίνονται, το Μαγεύσκι στην Πολωνία και ε, άλλη μία στην Αυστρία γίνονται πιο αναπτυγμένες περιοχές. Αυτό για να σας δείξω ότι έχουν αλλάξει στοιχεία. Η κεντρική Ελλάδα έχει στοιχεία 98% ε, ΑΕΠ επί του 2006-2008 ε, και 86% ε, επί τη βάση του μέσου όρου της Ευρώπης των 27, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία ΑΕΠ για το 2009. Το πρώτο μας μέλημα και ενδεχόμενη πρόταση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δει ποιε είναι οι επιλογές οι οποίες παρουσιάζονται σε αφορά αυτή την αστάθεια των στοιχείων. Ας πούμε, μια ενδιάμεση αναθεώρηση της επιλεξιμότητας για την επόμενη προγραμματική περίοδο και τον τρόπο με τον οποίο ενδεχομένως θα μπορούσε κανείς να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση. Μπορούμε βεβαίως να αναπτύξουμε περαιτέρω το θέμα αυτό αργότερα εάν ε, καταστεί απαραίτητο. Επίσης, βλέποντας τα στοιχεία οποία ε, προβληματιζόμαστε για τον τρόπο με τον οποίο προηγούμενες ε, περιοχές χρηματοδότησης ε, σύγκλησης ε, έχουν χρησιμοποιηθεί σαν βάση για την κατανομή των κονδυλίων. Δηλαδή η προηγούμενη επιλεξιμότητα είναι αυτή η οποία καθορίζει την κατανομή των κονδυλίων και όχι απαραίτητα η παρούσα κατάσταση και αυτό θα πρέπει ενδεχομένως να αναθεωρηθεί. Επίσης υπάρχουν και στοιχεία σαφή στην πρόταση της Επιτροπής, κυρίως τα κριτήρια για τις πιο αναπτυγμένες και τις υπομετάβαση ε, περιο περιφέρειες. Ε, επίσης όσον αφορά την ε, διάρθρωση του προπολογισμού και την επίπτωση που θα μπορούσαν να έχουν στον προπολογισμό των διαφόρων χωρών καθώς επίσης και την, τα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με το κάπινγκ καθώς επίσης και με, την, με, τον αντιστραμμένο, με την συγκεκριμένη σύγκληση. Όσον αφορά τώρα τους ε, ε, την, ε, τις πράσινες πολιτικές νομίζω ότι βλέπουμε να υπάρχει ευρεία συνέχιση τουλάχιστον στους στρατηγικούς στόχους, σε επίπεδο στρατηγικών στόχων και όσον αφορά βεβαίως και την εδαφική συνοχή. Υπήρξε φυσικά και η ε, μεταστροφή προς το πρόγραμμα της Ευρώπης 2020 ε, καθώς επίσης ε, και η κατάτμιση της αρχιτεκτονικής αυτής σε δύο μεγάλους στόχους. Το κύριο μέλημά μας εδώ είναι η έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τους αντικειμενικούς στόχους. Κυρίως από την πλευρά που το βλέπουμε εμείς τουλάχιστον η διαφορά ανάμεσα στους στόχους ε, Ευρώπης 2020 και τους στόχους της συνοχής. Προτείνομαι να υπάρξει ένα νέο άρθρο για τους ε, στόχους ε, έτσι ώστε στις πρόνοιες του κανονισμού να αποσαφηνίζονται και οι πρωτοβάθμοι και οι δευτεροβάθμοι στόχοι. Εναλλακτικά, στο άρθρο 2 θα μπορούσαν να γίνουν τα πράγματα πιο σαφή, εκεί που αναφέρονται δηλαδή οι όροι. Ε, και... Ε, και οι ορισμοί. Ε, αυτά τα ζητήματα, εάν διευθετηθούν, οπωσδήποτε θα προσθέσουν πολύ μεγαλύτερη ε, σαφήνεια για τους στόχους της επόμενης προγραμματικής περίοδου. Ένα άλλο σημαντικό θέμα ε, που συνδέεται με την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης ε, ε, είναι η εδαφική διάσταση. Αυτό γίνεται σαφέστερο στο προσχέδιο του κανονισμού, κυρίως δε στο σημείο της ενδυνάμωσης της τοπικής ατζέντας. Ε, γίνονται προτάσεις ε, σχετικά με επενδύσεις ε, αηφόρου ανάπτυξης, ολοκληρωμένες επενδύσεις κτλ μας απασχολεί αυτή ε, η ανάλυση top-down ε, των περισσότερων ε, θεμάτων, καθώς επίσης και η έλλειψη συγκεκριμένων βημάτων για την οικοδόμηση ικανοτήτων. Πιστεύουμε ότι μεγαλύτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στα τοπικά και περιφερειακά εδαφικά εργαλεία, τα οποία μπορούν να προηθηθούν και από τα κράτη-μέλη. Βλέπουμε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στην αστική ανάπτυξη ε, ενδεχομένως μπορεί βεβαίως ε, να αναθεωρηθεί και να επαναδιαπραγματευτεί το ring fencing ε, και επίσης θα μπορούσε να γίνει πιο ενδεικτική η παρουσία των πόλεων αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά τα θέματα είναι θέματα άλλωστε τα οποία έθιξε και ο Νίκολας Μάρτιν χτες. Μας απασχολεί επίσης ε, το επίπεδο ε, ικανότητας ε, το οποίο θα πρέπει να προϋπάρχει έτσι ώστε να εφαρμοστούν κοινοτικά κεντρικά προγραμματισμένα προγράμματα. Ο προβληματισμός μας προέρχεται ή μάλλον απορρέει από προηγούμενα προγράμματα τα οποία είχαν εστιαστεί στην αξιολόγηση εξάντε για διακρύβωση του κατά πόσον ε, ε, υπάρχει, υφίσταται η ικανότητα. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει πάντα, ελοχεύει σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος απώλειας ε, της στρατηγικής κεντρικής, ας πούμε, του στρατηγικού κεντρικού σχεδιασμού. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ε, στο CSF, ε, κυρίως δε στην εδαφική διάσταση, ένα πιο συγκεκριμένο κεφάλαιο ή να ενδυναμωθεί το υπάρχον κεφάλαιο, ε, ενδεχομένως παίρνοντας το σημείο αναφορά στην Ατζέντα 2020 και να συμπεριλαμβάνεται και ένα ιδιαίτερο τμήμα στα παραρτήματα ή στο παράρτημα που θα αναφέρεται στην εδαφική συνοχή, ε, όπου θα αναφέρεται με ποιο τρόπο μπορεί να ληφθεί υπόψη αυτή η εδαφική συνοχή ε, στα πλαίσια των θεματικών ε, πρωτοβουλειών, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η εδαφική πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη, ας πούμε, την εδαφική συνοχή, καθώς επίσης και τις δυνατότητες και τη δυναμική που παρουσιάζει η κάθε περιφέρεια Επίσης όσον αφορά την ε, ε, εδαφική συνεργασία θεωρούμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να είμαστε πιο συγκεκριμένοι έτσι ώστε να είναι, αποτελεσματικά και, να είναι αποτελεσματική και αυτή, η, αυτός ο συντονισμός, αυτή η συνεργασία και επίσης η συνεργασία αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να συνάδει με ένα βαθμό ε, συμπίκνωσης ε, το οποίο θα πρέπει να ε, μπορεί να προβλεφθεί και που θα πρέπει να αποτελέσει μία από τις προτεραιότητες ή εν πάση περιπτώσει να μειωθεί το ποσοστό των, των πρωτοβουλειών. Θα πρέπει να υπάρξει κάποιος μηχανισμός συντονισμού ανάμεσα στα συμβαλόμενα ε, από πλευρά των διαφόρων ε, ε, κρατών. Ενδεχομένως να υπάρξει ένα μνημόνιο κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, λαμβάνοντας υπόψη και τις μακροοικονομικές και τις μακροπεριφερειακές πολιτικής. τώρα θα, αφήσω, θα δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου Κάρλος Μέντες για την παρουσίαση του υπόλοιπου κομματιού. Ευχαριστώ. Έρχομαι στη στρατηγική συνοχή και τον προγραμματισμό. Το έχουμε ήδη εξετάσει λεπτομερία στη προηγούμενη έκθεση, αλλά τώρα εκτός από την εδαφική διάσταση, το θέμα είναι πώς θα εγκριθεί αυτό το έγγραφο. Συμφωνούμε με την αίσθηση του Κοινοβουλίου και πολλών κρατών μελών ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχουν νομοθετικό ρόλο να διαδραματίσουν εδώ και τα άλλα θεσμικά όργανα, Επιτροπή Περιφερειών βεβαίω και Κοινωνική Επιτροπή και Οικονομική να συμμετέχουν ε, στη διαβούλευση περισσότερο αντί να είναι κατεξουσιοδότηση πράξη ε, για τι συμβάσει εταιρική σχέση συμφωνίες όπως ε, ονομάζονται και τα επιχειρησιακά σχέδια και προγράμματα. Κατά πρώτο και κύριο λόγο, εμείς πιστεύουμε ότι η εδαφική συνοχή και οι στόχοι της θα πρέπει να αντανακλώνται σαφώς στο περιεχόμενο αυτών των εγγράφων. Διαβάζοντα το σχέδιο κανονισμού δεν έχει κανείς αυτή την αίσθηση αμέσω ω προς το περιεχόμενο του. Η εδαφική διάσταση μπορεί να αναφέρεται, αλλά στην πλευρά τη ενσωμάτωση και τη ολοκλήρωση. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πραγματικά να είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, όχι συμπληρωματική και μια ήπια μορφή συντονισμού, εν περιπτώσει, αλλά πλήρης ένταξη ε, με συνέργειες, ε, με προγράμματα από πολλαπλή χρηματοδότηση από διάφορα ταμεία. Υπάρχει αυτή η ιδέα βεβαίως ε, επιλεκτικά ε, με ε, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και το Κοινωνικό Ταμείο. Προαιρετικά, τουλάχιστον στη Σκωτία υπάρχει αυτή η δυνατότητα ε, να μπορούμε να τρέχουμε σε αυτά τα ταμεία αυξημένη διασταυρούμενη χρηματοδότηση, το 5%. Βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν περίπλοκες καταστάσεις εκεί, αλλά τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες θα μπορούσαν προαιρετικά και πάλι να επιλέγουν αν θέλουν να έχουν ψηλότερο κατόφλι. Επίσης, υπάρχει και κάποια έλλειψη συνοχής ε, οι επενδυτικές προτεραιότητες ε, στο Περιφερειακό Ταμείο, ενώ δεν είναι σε άλλα ταμεία προτεραιότητα. Για το Κοινοβούλιο μπορεί να μην είναι μεγάλη προτεραιότητα κάτι άλλο. Για το Συμβούλιο μπορεί να είναι, αλλά οι βασικές ανησυχίες των ε, συμβάσεων εταιρικής σχέσης και των προγραμμάτων ε, δεν θα πρέπει να επικαλύπτονται μάλλον αυτά τα δύο. Αυτή είναι η βασική ανησυχία. Και η Επιτροπή κάνει μια πρόταση όπου το πεδίο εφαρμογή δεν είναι αρκετά μεγάλο. Είναι πιο περιοριστικά, πιο δεσμευτικά ε, αυτά που προτείνει από κάποιες άλλες στρατηγικές. Τώρα για τη θεματική συγκέντρωση ή την οριοθέτηση, αυτό το ring fencing, ο καθένα θα συμφωνήσει ε, καταρχήν για τη συγκέντρωση σε συγκεκριμένε θεματικέ ενότητες, αλλά μετά τα κράτη-μέλη, περιφέρειες ε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αντίθετα προ τις προτάσεις αυτές. Εμεί την προτείνουμε. Να χρειάζεται αιτιολόγηση για αυξημένη συγκέντρωση σε κάποια προγράμματα και εκ των προτέρων ε, εκτίμηση Δηλαδή αν υπάρχει αύξηση να αιτιολογείται και να αποδεικνύεται ότι αυτό θα βοηθήσει για να επιτευχθεί μια κρίσιμη μάζα. Το ίδιο ισχύει και για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Δηλαδή, αντί να έχουμε ε, τεχνητούς ε, και πολύ αυθαίρετους στόχους εκ των προτέρων, θα πρέπει να είναι οι ανάγκες ε, της περιφέρειας εδαφικές που να ορίζουν και οι δυνατότητες απορρόφησης και σε συνεργασία με όλους ενεχομένους τι θα ισχύει. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν θα πρέπει να αυξήσει τους πόρους. Μπορεί να χρειαστεί να τους αυξήσει, αλλά να υπάρχει αποχρόν λόγος για κάθε χώρα μέλος και για κάθε περιφέρεια. Το πλαίσιο επιδόσεων τώρα, η αιρεσιμότητα συζητήθηκε πολύ εδώ στο Κοινοβούλιο και στην περασμένη έκθεση συμφωνήσαμε ε, εκ των προτέρων αιρεσιμότητα να υπάρχει εξάντεν. Υπάρχουν και κάποιες γενικές ε, συνθήκες και όροι που ε, συμμορφούνται με κάποιες άλλες πολιτικές της Ένωσης και επίσης η λεγόμενη μακροοικονομική αιρεσιμότητα νομίζουμε ότι είναι νομικά αφιλεγόμενη αυτή η υπόθεση και αμφίβολη. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει συνταγματική βάση. Είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση από το Ταμείο Συνοχής, το οποίο ήρθε το 1993 και συνδέθηκε ρητά με τα κριτήρια σύγκλησης και την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης το Κοινωνικό Ταμείο δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Το πλαίσιο επιδόσεων λοιπόν δεν θα πρέπει να είναι ένα αποθεματικό ε, που να απορροφά κονδύλια. Θα πρέπει να συνδέεται με αποτέλεσμα, να, οι δείκτες να είναι αποτελέσματος και όχι οι οικονομικοί δείκτες και, output. Το ελεκτικό συνέδριο το επισήμανε πέρυσι. Ε, συγγνώμη, τον περασμένο μήνα και θα πρέπει να υπάρχει αξιόπιστη και πληροφόρηση και σωστή μεθοδολογία, επίσης αξιόπιστη. Γενικά συμφωνούμε με την εξάντε αιρεσιμότητα για τα στατιστικά συστήματα και τους δείκτες αποτελεσμάτων Κοινού δείκτε επίση χρειαζόμαστε. Ξέρω ότι γίνεται συζήτηση κατά πόσο θα πρέπει αυτό να μπει στον κανονισμό ή κάπου αλλού, σε κάποιο άλλο έγγραφο. Για μα αυτό που έχει σημασία είναι να ε, έχουν συμφωνηθεί στην αρχή τη προγραμματική περίοδου και όχι κατά τη διάρκεια τη. Και επίση να υπάρχει κάποια συνέπεια και συνέχεια έτσι ώστε ο κανονισμό του Ταμείου Περιφερειακή Ανάπτυξη να μην διαφέρει από κάποιου άλλου δείκτες αποτελέσματο, παρόλο που αναφέρονται να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι δείκτε αποτελέσματο, γιατί και πάλι δημιουργείται σύγχυση στις διαχειριστικές αρχές, τους φορεί. Το βλέπουμε στις εκθέσεις υλοποίησης. Μια καλή αρχή θα ήταν να τα ρυθμίζουν αυτά τα νομικά κείμενα από την αρχή και να διατηρείται κάποια συνέπεια σε όλα τα ταμεία και μια συνοχή. Επίσης θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι όσο γίνεται μεγαλύτερη πρόσβαση ε, για την αξιολόγηση όπως λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα σας δώσω ένα παράδειγμα αργότερα προς την ε, Κομισιόν. Ε, τη δυνατότητα τώρα είναι πολύ ε, σημαντική η μεγαλύτερη εστίαση και την καλωσορίζουμε, αλλά χρειάζονται και δείκτες για συγκριτική αξιολόγηση, benchmarking δηλαδή. Το, τα σχέδια κοινή δράση βεβαίω τα υποστηρίζουμε. Είναι χρήσιμο ω μια δοκιμή και θα μπορούσε ενδεχομένω στο μέλλον αυτό να γενικευθεί και σε άλλα προγράμματα και σε όλα τα ταμεία. Ένας τομέας που νομίζουμε ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα και έλλειμμα είναι το θέμα της λογοδοσίας. Ακούσαμε πολλά εδώ για πολιτική συζήτηση υψηλού επίπεδου ε, στη έκθεση συνοχής και μέχρι να έρθει νομοθετική πρόταση ε, και σε άλλες εκθέσεις, αλλά στη νομοθετική πρόταση δεν γίνεται μεγάλος λόγος. Προτείνουμε ένα πλαίσιο ε, λογοδοσίας της ε, επίδοσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια ετήσια ε, μορφή έκθεσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο και θα επανέλθω σε αυτό, ετήσια συζήτηση στο Συμβούλιο. Τουλάχιστον δεν υπάρχει βούληση για σχηματισμό ειδικό του Συμβουλίου που να ασχολείται με αυτά τα θέματα. η αξιολόγηση μεταξύ ομοτήμων σε ένα νέο ε, είδος ε, ομάδας εργασίας υψηλού επίπεδου και για να υποστηριχθεί όλο αυτό το πλαίσιο επιδόσεων θα πρέπει και οι εκθέσεις υλοποίησης και ιδίως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και του προγράμματος να εστιάζονται ακριβώς στα αποτελέσματα. Όχι απλώς κατά πόσο υπάρχει απορρόφηση των χρημάτων και λειτουργικά στοιχεία. Ένα κεφάλαιο για τις επιδόσεις λοιπόν θα μπορούσε να ενταχθεί στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να είναι και η βάση μάλιστα για μια τέτοια έκθεση επιδόσεων και προτείνουμε να σβηστούν πολλές λεπτομέρειες που υπάρχουν σήμερα στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι όλα αυτά μπαίνουν στην έκθεση πεπραγμένων την ετήσια με τρόπο πιο λεπτομερή και αναλυτικό, οπότε δεν χρειάζεται αυτή η επικάλυψη. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα αποτελέσματα και όχι δείκτες οικονομικής ε, απορρόφησης ή output. Το ίδιο ισχύει και για τα κείμενα και τις εκθέσεις ε, υλοποίησης των προγραμμάτων. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ενίσχυση των ελάχιστων προδιαγραφών στο μοντέλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίσης να δημοσιεύονται στο σύνολό τους μέχρι τον Ιούνιο του επομένου έτους, το αργότερο. Όχι μια σύνοψη για τους πολίτες, η πλήρης έκθεση να δημοσιεύεται με τις επιδόσεις όσο γίνεται νωρίτερα τον Ιούνιο δηλαδή του επομένου έτους. Και στην τελευταία διαφάνεια για την απλοποίηση και την ε, αξιοπιστία συμφωνούμε σε πολλά από αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επειδή δεν έχω και χρόνο βλέπετε στη διαφάνεια ποιο είναι το πιο σημαντικό αξιολόγηση να είναι συστηματική ε, αναθεώρηση των προτάσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε κάποιες μελέτες Υπάρχει ένα κόστος της μεταρρύθμισης, αλλά θα πρέπει το συντομότερο να ενημερωθεί το Κοινοβούλιο για αυτή τη μελέτη, για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Εμείς θεωρούμε ότι η βασική προτεραιότητα είναι απλοποίηση για τη διαχειριστική αρχή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχυρίζεται ότι η προτεραιότητα είναι για τους δικαιούχους. Και επίσης η απλοποίηση, η απλούστευση να είναι βασικό χαρακτηριστικό του νέου πλαισίου επιδόσεων και ε, λογοδοσία. συμπεριλαμβανομένων και των μελετών που αναθέτει εκ των υστέρων Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο για τα μέτρα απλοποίηση κατά τη διάρκεια της περίοδου και να ελέγχονται αυτά και περιοδικά να αναφέρονται στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ. Θα οδηγηθούμε γρήγορα στον κύριο Σούλε και ε, θα του διαθέσουμε 10 λεπτά. Ευχαριστώ. Περιμένω να αρχίσουν οι διαφανίες μου. Ευχαριστώ και πάλι όμως που με καλέσατε. Είναι δύσκολο να ε, προχωρήσει κανείς μετά από μία τόσο συνεκτική παρουσίαση και αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω είναι να παρουσιάσω τη στρατηγική κατεύθυνση ε, στην οποία βλέπω ότι πρέπει να διατυπωθούν οι προτάσεις. Θέλω να σας πω ότι εργαζόμαστε για το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής που είναι ένα think tank, ε, ένα όμιλος περισυλλογής και ε, ε, εξετάζουμε το πολιετές πλαίσιο, έχουμε ε, δημοσιεύσει διάφορες σκέψεις και θα κάνω ορισμένα σχόλια τα οποία μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα μας. Υπάρχει όμως μία αναφορά εδώ η οποία τονίζει και αποβλέπει στην απλοποίηση πού οδηγείται η περιφερειακή πολιτική. Καταρχήν συμφωνώ με τους στόχους που έχουν καταρτιστεί, τους γενικούς στόχους, τους οποίους έχω καταγράψει εδώ, η Ευρώπη του 2020 προσανατολίζεται για αποτελέσματα, χρειάζεται ε, μία ολοκληρωμένη προσέγγιση, απλοποίηση στη χρήση των πόρων για να υπάρχει και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Όλα αυτά ωραία ακούγονται, αλλά πώς ερμηνεύονται στην πρακτική διότι έχω ξαναεξετάσει προηγούμενα πολυετή προγράμματα πλαίσιο και ουσιαστικά βλέπουμε ότι οι ίδιοι όροι χρησιμοποιούνται και τότε. Αλλά δεν είχαμε πάντοτε τη σωστή εφαρμογή. Αυτό που είναι σημαντικό και πρέπει να τονιστεί είναι ότι υπάρχει μία επιμονή των αντιφάσεων που είναι κάτι το αναπόφευκτο. Το θέμα είναι τι θέλετε να τονίσετε περισσότερο, τι λιγότερο και δεν υπάρχει και μία σαφής ε, ε, στρατηγική ως προς την κατεύθυνση. Οι πόροι χρησιμοποιούνται για όλα, πρέπει να καλύψουν τα πάντα συγχρόνως και αυτό δημιουργεί ορισμένες αντιφάσεις στη λειτουργία τους. Θα ε, αναφερθώ σε ορισμένες από Καταρχήν, πόσο ε, περιφερειακή θα είναι η περιφερειακή πολιτική. Ε, θα χρειαστεί να υπάρχει συνεκτικότητα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, με το πρόγραμμα Ευρώπη το 2020 και θα πρέπει να υπάρχει και μία σαφής ε, εφαρμογή. Οι συμφωνίες ε, ε, συνεργασίας οι οποίες είναι κάτι από τα θέματα που είναι πολύ επίκαιρα πώς θα τις διαπραγματευτούμε και μπορεί να υπάρχει διαφορά στην αντιμετώπιση τους ανάμεσα στα κράτη-μέλη οπότε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα στη συνέχεια. Επίσης θα πρέπει ε, να υπάρχει ε, μία κατεύθυνση η οποία θα δοθεί από την περιφέρεια στο θέμα αυτό. Ε, όσον αφορά την θέση μεταξύ της θεματικής συγκεντρώσεως και των συμβάσεων συνεργασία γιατί έχουμε και τα δύο διότι εάν οι συμφωνίες συνεργασίες πρόκειται να μας δώσουν το πλαίσιο στο οποίο θα υπάρξει η ανάπτυξη γιατί να έχουμε και τις θεματικές συγκεντρώσεις. Οι περιφέρειες θα μπορούσαν να καθορίσουν ποιες είναι οι περιοχές στις οποίες θέλουν να επενδύσουν, που έχουν τα μεγαλύτερα κενά και δεν χρειάζεται να υπάρχει αυτή η θεματική συγκέντρωση. Όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση, ε, επηρεάζει τις πολιτικές ε, μήπως υπάρχει μία πιο καθευθυντική ε, προσέγγιση ε, και ποια θα πρέπει να είναι η μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση. Όσον αφορά το θέμα της απλοποίησεως, δεν θέλω εδώ να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Πάντοτε προσπάθησαν να απλοποιήσουν τα προγράμματα, αλλά το πρόβλημα είναι η εφαρμογή, η οποία σημαίνει ότι χρυσώνουμε το χάπι και στο τέλος όταν δούμε την πρακτική εφαρμογή στην περιφέρεια η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Επίσης τι επιτρέπεται βάσει των κανόνων ανταγωνισμού. Όλα αυτά τα οποία ζητούνται είναι απαραίτητα και όσον αφορά την μελλοντική συνεργασία υπάρχει δυνατότητα μέσω αυτών των ε, διαπραγματεύσεων να υπάρξει ε, μία ε, προσέγγιση αποφυγής των κινδύνων. Δηλαδή αντί να ξεκινήσει κανείς από τα λίγα προς τα πολλά να χρησιμοποιηθεί η αντίθετη πορεία το οποίο αποτελεί επίσης ένα κίνδυνο προς αποφυγή υπερβάσεων. Έχουμε και ένα ερώτημα που αναφερόταν στις διάφορες περιοχές. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των περιφερειών, υπάρχει και διαφορετική θεματική συγκέντρωση και διαφορετική χρηματοδότηση και η διαφορά που πρέπει να μας απασχαλήσει ε, όσον αφορά τις περιφέρειες και τις ε, διαφορές τους αρνητικά είναι ότι υπάρχουν ορισμένες ε, περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση στην ισχύουσα χρηματοδότηση ενώ θα υπάρξουν ε, νέες ροές χρηματοδοτήσεων και είναι δύσκολο να δούμε πώς οι περιφέρειες θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις νέες δυνατότητες αν δεν έχουν πολύ ανεπτυγμένη διοικητική δυνατότητα και υπάρχουν ε, περιοχές οι οποίες ε, ε, πηγαίνουν καλύτερα, άλλες οι οποίες πηγαίνουν χειρότερα και πρέπει να ληφθεί και αυτό υπόψη. Η αιρεσιμότητα, η το απόθεμα αποδόσεως. Όταν όλα αυτά συνδυάζονται με χρηματοδότηση πρέπει κανείς ε, ναι ε, να ε, εκπληρώνει τις προϋποθέσεις και να κοιτάξει να πάρει ε, την ε, χρηματοδότηση μετά όμως ε, αυξάνεται η γραφειοκρατία αντί για το αποτέλεσμα. Υπάρχουν βέβαια και ορισμένοι οι οποίοι τα καταφέρνουν σε μια περιφέρεια εάν πηγαίνει καλά η περιφέρεια μπορεί να μην επηρεαστεί από την κατάσταση του κράτους μέλους. Δεν είναι προφανές αλλά αυτό, τέτοια παραδείγματα έχουμε δει ήδη. Ένα άλλο θέμα που δεν έχουμε εξετάσει επαρκώς στις ε, ε, μεταρρυθμίσεις είναι η επίπτωση της κρίσης και ιδίως της κρίσης στην Ευρωζώνη και βλέπουμε ότι ε, αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους έχουμε μία τάση για τη συνέχιση της κρίσεως στην Ευρωζώνη και πρέπει να ξανασκεφτούμε πόσο θα ε, ε, δαπανίσουμε αυτή τη χρηματοδότηση διότι διαφορετικά μπορεί να μην χρειάζεται αλλά αν κοιτάξουμε την συνεχιζόμενη διαρθρωτική κρίση ίσως πρέπει να δούμε ε, τι, πώς θα πορευτούμε διότι πρέπει να δούμε το ΑΕΠ κατά κεφαλή αλλά κοιτάζουμε την διαφορά σε αποδοτικότητα, βλέπουμε τα προβλήματα που υπάρχουν σε ορισμένες χώρες, διότι υπάρχουν ή ε, στην ε, χρηματοδότηση συνοχής δυνατότητες, αλλά μπορούμε να προεξοφλήσουμε ότι οι κανόνες ισχύουν στις περιοχές αυτές και τι πρέπει να στηρίξουμε περισσότερο. Έναν μηχανισμό μηχανισμό μεταφοράς, ένα μηχανισμό συνοχής για στήριξη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή περισσότερες δαπάνες. Έχω ακόμη 30 δευτερόλεπτα, οπότε προσπάθησα να σεβαστώ το χρόνο μου. Πολλά από τα μέτρα είναι στη σωστή κατεύθυνση, αποτελούν καλές καινοτομίες, ε, είναι καλές οι προτάσεις, αλλά υπάρχει όλο και περισσότερο μία ε, κίνηση για ε, έλεγχο ε, εκ των άνω προς τα κάτω ε, και υπάρχει το θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης. Πολλά εξαρτούνται από την απλοποίηση η οποία στο χαρτί δεν σημαίνει υποχρεωτικά και στην ουσία απλοποίηση. Υπάρχουν και πολλές αλλαγές οι οποίες οδηγούν σε επιπλέον ανασφάλεια ε, και σε μία κάλυψη, συγκάλυψη των ατελειών. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει τουλάχιστον ένα ελάχιστο περιθώριο συμμορφώσεως και όχι ένα μέγιστο. Γενικώ πιστεύω ότι η στρατηγική αυτή η κατεύθυνση του Ταμείου δεν έχει αλλάξει και ολοκληρώνω λέγοντας ότι η πραγματική επίπτωση των αλλαγών είναι για ε, τις, ε, τα μέτρα αυτά τα οποία θετικά, όχι όμως αρκετά προοδευτικά. Ε, δεν χρειάζεται να σχολιάσω τις λεπτομέρειες. Ποια θα είναι η διαφορά μεταξύ των κρατών μελών είναι κάτι που παραμένει ακόμη προς συζήτηση και τέλος πρέπει να δούμε τι θα γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να μπορέσουμε να προωθήσουμε ε, την στήριξη ιδίως στις περιοχές που δεν μπορούν μόνες τους να τα βγάλουν πέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον επόμενο ε, ομιλητή μας, εμπειρογνώμονα, ο κύριος Μάρκους Τρίλινγκ ε, ο οποίος είναι από το Bank Watch. Μπορείτε να πείτε αν θέλετε κάτι για τον εαυτό σας. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Μάρκος Τρίλινγκ. Ευχαριστούμε για την δυνατότητα που μας δίνεται σήμερα ε, να ασχοληθούμε με τους δείκτες και την αξιολόγησή του. Σήμερα το πρωί ε, η κυρία Χέντεγκαρντ ασχολήθηκε με το θέμα αυτό και ο κύριος Όλμπρεχτ αναφέρθηκε στο θέμα, στο ίδιο θέμα και θα ήθελα να σας δείξω ε, κάπως ε, ε, τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να ειδωθούν αυτοί οι δείκτες και βάσει του πλαισίου του, της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ξεκινώντας από τη συγκέντρωση των πόρων, την ε, απλούστευση από τα χαρτιά στην πραγματική ε, απόδοση και πρέπει να πω μάλλον ότι ε, ο στόχος του αποτελέσματος πρέπει να οδηγήσει σε μία διαφορά προσέγγισης. Έχουμε και σχόλια άλλωστε από το ελεγκτικό συνέδριο προς την ίδια, κατάστα... προς την ίδια κατεύθυνση την οποία ελπίζω ότι θα μπορέσω να σας δείξω. στο ερώτημα πώς μπορεί να ε, ε, καθιερωθεί ο δείκτης αποτελέσματος ε, στην οδηγία το, το συνέδριο αναφέρει ότι ακόμα αυτός ο δείκτης αφορά ε, μάλλον τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς και όχι την απόδοση. Και θα πρέπει ε, να οδηγηθούμε ε, ακριβώς στους λεγόμενους result indicators, δείκτες αποτελέσματος, που θα αφορούν ακριβώς το αποτέλεσμα και την απόδοση και όχι μονάχα τη συμμόρφωση. Έχουμε επίσης ε, και το συγκεκριμένο έτοιμα ε, της 17ης όπου αναφέρεται ακριβώς εις ε, την, στις επίσημες απαιτήσεις σε σχέση κυρίως με τους θεματικούς στόχους ή προτεραιότητες και ε, βάσει αυτού θα πρέπει να δίδονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο, τον συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο ε, ε, τα κονδύλια συμμετέχουν στην βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης του πληθυσμού. Μιλάμε για στόχους, μιλάμε για στοχοθέτηση. Όποιος μιλάει για στόχους βεβαίως ε, θα πρέπει να έχει και κάποιους δείκτες έτσι ώστε να καταδεικνύεται κατά πόσον και μέχρι ποιο βαθμό έχει επιτύχει το στόχο του. Εδώ έχουμε ε, τους στόχους της Ευρώπης 2020, ε, έχουμε επίσης ε, και την, τους στόχους υφόρου ανάπτυξης και το, κεκτημένο, το περιβαλλοντικό κεκτημένο που θα πρέπει να καλυφθούν βεβαίως. Η δεύτερη λειτουργία είναι ακριβώς ε, οι δείκτες που θα πρέπει να μας δείξουν πώς, ε, το κατά πόσον ε, υπάρχει πρόοδος και το βαθμό στον οποίο θα έχουμε επιτύχει τους στόχους μας και βεβαίως στο τέλος θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε την εφαρμογή της πολιτικής και το κατά πόσον έχει πετύχει ή όχι. Κοινοί δείκτες έτσι όπως εμφανίζονται στον κανονισμό ενδεχομένως ε, μπορεί να έχουν τα χαρακτηριστικά ε, του output indicator έτσι όπως τον ε, θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ βλέπουμε ας πούμε τον αριθμό των επιχειρήσεων που μπορούν να συμμετέχουν, τον αριθμό των επιχειρήσεων που λαμβάνουν άλλες επιδοτήσεις κτλ αυτοί οι προτινόμενοι κοινοί ε, δείκτες τελικά δεν αποτελούν ε, ικανοποιητικό και αρκετό ε, τρόπο διασύνδεσης με, την Ευρώπη, με τους στόχους της Ευρώπης 2020, ούτε βελτιώνουν την ποιότητα του στόχου πολύ συχνά απλώς έχουν περιγραφικό χαρακτήρα, επομένως χρειάζεται monitoring, χρειάζεται τακτική επιθεώρηση ενδιάμεσες επιθεωρήσεις. Και τέλος υπάρχουν και ήδη και κάποια πολύ καλά παραδείγματα ε, στη Σλοβεκία και σε άλλες ε, χώρες ε, όπου έχουν χρησιμοποιηθεί πιο εξεζητημένοι δείκτες. Αυτό που θέλω να προτείνω εδώ είναι μία σειρά δικτών που θα τους ονομάσω ε, ε, περιφερειακούς, ε, συγγνώμη, δείκτες αηφόρου περιφερειακής ανάπτυξης. Πρέπει να πω βεβαίως ότι και όλοι οι δείκτες οι οποίοι αναφέρονται εδώ βεβαίως είναι διαθέσιμοι τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο και ότι τελικά βεβαίως ο όγκος είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτό που παρουσιάζουμε εδώ. Επίσης όταν μιλάμε για καινοτομία, τεχνολογική ανάπτυξη ε, και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν δείκτες ε, οι οποίοι είναι σημαντικοί και οι οποίοι ε, δείχνουν τι σημαίνει μέχρι που έχει φτάσει το πρόγραμμα στις επιχειρήσεις και βεβαίως και το θέμα της ε, ανταγωνιστικότητας και της ε, περιβαλλοντικής πολιτικής, δηλαδή σε σχέση με το κλίμα και τα λοιπά, όλα αυτά τα στοιχεία ε, είναι, επίσης υπάρχουν στοιχεία σχετικά και δείκτες σχετικά με την ενεργειακή ένταση και τα λοιπά είναι όλοι δείκτες που επηρεάζουν την οικονομία μας. Υπάρχουν επίσης δείκτες ε, που δείχνουν ανατομέα την εκπομπή αερίων θερμοκηπίου. Ε, στα πλαίσια της πολιτικής 2020 μιλάμε για ανανεώσιμες ε, ε, ενέργειες και βεβαίως υπάρχει δίκτυση σχετικά με το κομμάτι που το ρόλο που παίζουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο, στο τελικό ενεργειακό μείγμα. Έχουμε πληροφορίες επίσης σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την ικανότητα καινοτομίας. Ένας Άλλος ε, δείκτης ε, είναι των, ε, των πόρων και του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται έτσι ώστε ας πούμε να υπάρχει συγκεκριμένος δείκτης για την για την πραγματική κατανάλωση ανα νοικοκυριό και ανακάτοικο. κάτοικο. Ο, επίσης για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ηχορύπανσης και της ρύπανσης του περιβάλλοντος ε, στις πόλεις και ε, επίσης ε, τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να διασυνδέσουμε τη στέγαση με την ποιότητα ζωής ε, των πολιτών και για τις όσον αφορά τώρα την προώθηση αηφόρων τρόπων ε, μεταφοράς και τα για να σταματήσει να υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση και τα λοιπά ε, θα υπάρχουν δείκτες σχετικά με το model split των, ε, της μεταφοράς επιβατών αλλά και της μεταφοράς εμπορευμάτων. Οι δείκτες ε, λοιπόν μπορούν να είναι ένα εργαλείο μέτρησης των στόχων σε εθνικό επίπεδο. Βεβαίως, ένας ε, φιλόδοξος στόχος θα μπορούσε να είναι αυτός της ε, στρατηγικής 2020. Εγώ εδώ ας πούμε παρουσιάζω μία προτεραιότητα και την παρακολουθώ στα πλαίσια του στόχου του 2020 και μέχρι το 2022. Αναφερόμαστε στην οικονομία ε, με μικρή έκκληση διοξιδίου του άνθρακος. Είναι ο στόχος του 2020 ε, και μπορούμε λαμβάνοντας υπόψη κεντρικά ε, στοιχεία για συγκεκριμένες χρονικές στιγμές εδώ 2016-2018 μπορούμε να ε, δούμε ε, το κατά πόσον προσεγγίζεται ο στόχος καθώς επίσης και το πλαίσιο υπό το οποίο μπορεί να αξιολογηθεί η πολιτική συνοχή. Αυτά είχα να σας πω ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε ήδη ξεπεράσει κατά 20 λεπτά το το χρονοδιάγραμμά μας. Ε, θα δώσω τώρα τον λόγο στον κύριο Γκαρτζούλο. Έχετε και κάποιον εμπειρογνώμονα μαζί σας νομίζω. Ε, σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την ε, ε, ευγενή σας πρόκληση, πρόσκληση, συγγνώμη, πρόσκληση, καθώς επίσης και για την ε, σημασία που δώσατε και στην περιοχή που εκπροσωπώ, την Κατάνια στην περιοχή αυτή είχαμε ένα από τα πιο σημαντικά επιχειρησιακά προγράμματα ε, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ είχα και, μία, και ένα οπτικό υλικό, το οποίο δεν το βλέπω όμως εδώ. Α, το βλέπω τώρα. È stata più Ehm, in Campania e a Napoli. Ε, διορθώνομαι εκπρόσωπος της ε, Καμπάνια. Ε, εγώ λοιπόν ε, ανήκω στη διαχειριστική ε, αρχή της περιφέρειας της Καμπάνια και επομένως είμαι υπεύθυνος για την εφαρμογή επιτόπου των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια της ε, παρούσας οικονομικής κατάστασης που όλοι γνωρίζουν να έχουμε και εμείς σε οικονομική ε, κρίση που όμως πρέπει να πω ότι έχει ξεκινήσει ήδη από την αρχή της δεκαετίας του 2000 ε, και εν πάση περιπτώσει συνεχίζεται ακόμα. Υπήρξε μια σημαντική ανάκτηση των ευρωπαϊκών περιοχών στόχου 1 που αναπτύχθηκαν με ποσοστό μεγαλύτερο από το ε, μέσο ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, των 27. Ε, στην Ιταλία όμως διαπιστώσαμε και μία διαφορετική τάση είχαμε και αύξηση των πιο πλούσιων ε, περιοχών. Εγώ θα προσπαθήσω στα 10 λεπτά που έχω στη διάθεσή μου, θα προσπαθήσω, λέω, να μιλήσω μόνο με το στόμα και να μην χρησιμοποιώ τα χέρια μου, να μην μιλήσω και με τα χέρια μου όπως οι περισσότεροι Ιταλοί. Αλλά αν μου επιτρέπει η πρόεδρος θα κάνω και καμιά χειρονομία. Ε, λοιπόν, έχουμε στην ε, περιφέρειά μας ε, ε, κάποια εδάφη τα οποία αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα. έχουμε ένα δημογραφικό τσουνάμι με ανάπτυξη του, του, της τάξης του 0%. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή και επομένως πρέπει να αντιμετωπιστεί και αυτό. Εγώ θα κάνω πρώτα κάποιες γενικές παρατηρήσεις αναφερόμενος ε, και στα θετικά και στα αρνητικά στοιχεία τα οποία διαπιστώνουμε ως φορείς ε, ε, που δουλεύουν επί τόπου όσον αφορά τα θετικά στοιχεία της νομοθετικής δέσμης ε, ε, μέτρων, με μεγάλη χαρά βλέπουμε την ε, εναρμόνιση των κανόνων όσον αφορά τα ταμεία συνοχής και τις πολιτικές συνοχής. Με ικανοποίηση επίσης βλέπουμε κοινές, κοινούς κανόνες όσον αφορά τις προγραμματικές περιόδους και αυτή τη στιγμή πρέπει να πω ότι έχουμε περισσότερα εργαλεία περιφερειακού σχεδιασμού που όμως δεν συντονίζονται απολύτως μεταξύ τους. Ε, Επίσης, ε, όσον αφορά τον, τη διαχείριση των ε, προγραμμάτων και αυτό είναι σημαντικό και η δυνατότητα κατανομής των κονδυλίων κατά δύο τρίτα στην περιφέρεια και στις στους οργανισμούς ε, διαχείρισης και αυτό θεωρούμε ότι είναι θετικό στοιχείο όπως επίσης και η ενίσχυση της αρχής ε, της ε, αναλογικότητας και των ελέγχων βάσει του επίπεδου κινδύνου της χρηματοδότησης. Και αυτό θεωρούμε ότι είναι σημαντικό στοιχείο. Θα αναφερθώ αργότερα στο θέμα αυτό προς το τέλος όταν θα αναφερθώ ακριβώς στους ε, ε, εκ των ελέγχους όμως ε, πρέπει να πω ότι δεν μας δίνεται η δυνατότητα ε, με ταχύτητα να προωθήσουμε το λειτουργικό μας πρόγραμμα, το επιχειρησιακό μας μάλλον πρόγραμμα. Ένα άλλο στοιχείο ε, είναι η ικανοποιητική, η αποτελεσματική χρήση της πληροφόρησης, δηλαδή η θέσπιση κοινών δικτών βεβαίως κάνει πιο εύκολη την αναφορά το reporting σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι προηγουλαλήσαντες συνάδελφοι αναφέρθηκαν ε, στη, στο θέμα αυτό, στη δυνατότητα δηλαδή περαιτέρω μείωσης ε, των ετήσιων ε, εκθέσεων έτσι ώστε να υπάρχει λιγότερο διοικητικό άχθος εις βάρος της, της, αρχής, της διαχειριστικής αρχής. Επίσης βλέπουμε ότι ε, αυτή η γενικότερη μείωση του διοικητικού άχθους ε, είναι κάτι θετικό. Θα πρέπει να ε, συνεχίσουμε τις προσπάθειες όσον αφορά τη λεγόμενη οικοδόμηση ικανοτήτων, capacity building των διαφόρων διοικήσεων. Ένα άλλο αρνητικό στοιχείο είναι η μείωση ε, το, του ε, διοικητικού κόστους εις βάρος των ε, δικαιούχων. Αυτή η νομοθετική δέσμη μέτρων υπογραμμίζει ιδιαιτέρως τον ρόλο των δικαιούχων. Κατά αυτήν την έννοια πιστεύω ότι η γραμμή που ακολουθείτε είναι ορθή. Θα αναφερθώ εντάχει στα αρνητικά Αυτά που πιστεύουμε ότι μπορεί να έχουν δηλαδή αρνητική επίπτωση στις διοικήσεις οι οποίες άμεσα καλούνται να διαχειριστούν τα τα ταμεία όπως ας πούμε αυτό το σύστημα των μακροοικονομικών ε, και του συστήματος ερεσιμότητας εξάντε. Το σύστημα αυτό ε, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα δημιουργήσει, θα προκαλέσει προβλήματα εάν δεν εφαρμοστεί ταυτοχρόνως ένα κριτήριο αναλογικότητας στην εφαρμογή του. Ε, ε, κυρίως φοβούμεθα ότι το κριτήριο ε, της αιρεσιμότητας θα πρέπει να εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο. Όσον αφορά τώρα και αναφέρομαι πάντα στα αρνητικά, ε, το πλαίσιο ε, αναφοράς ε, των αποτελεσμάτων και των προϋποθέσεων για την άρση των πόρων η διαδικασία διακρύβωσης επαλήθευσης θα πρέπει να απλουστευτεί κατά την άποψή μου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεκινήσει ευρεία συζήτηση ε, όχι μόνο με τους εμπλεκόμενους εθνικούς φορείς αλλά και τους ε, περιφερειακούς ε, φορείς που καλούνται, όπως έλεγα και προηγουμένως, να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού. Και το θέμα της εθνικής πιστοποίησης είναι κρίσιμη σημασίας κατά την άποψή μας όσον αφορά δηλαδή ακριβώς σε την διασφάλιση εξάντε. Ένα άλλο αρνητικό στοιχείο ή μάλλον όχι, επικριτικό, όχι αρνητικό ακριβώς, είναι το σύστημα ε, των ε, ε, ετήσιων λογαριασμών που πρέπει να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η υποχρέωση ετήσιου κλεισίματος ε, δαπανών ενδεχομένως θα δημιουργήσει προβλήματα, ε, όπως επίσης ε, και τα, τα συστήματα των ετήσιων λογαριασμών τα οποία θα πρέπει να φτάνουν μέχρι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφενός θα δυσκολέψουν την κατάσταση, αφετέρου καθόλου δεν θα την απλουστεύσουν γιατί βεβαίως η ανάγκη ε, για ε, έλεγχο των ε, λογαριασμών μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ενδεχομένως να δημιουργηθεί ένα είδος επικάλυψης ελέγχου των λογαριασμών γιατί μπορεί να γίνεται και από το Ελεγκτικό Συνέδριο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από τους, από από τους κατατόπους ελεγκτές. Ε, και το λέω γνωρίζοντα πάρα πολύ καλά, ε, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή διαχειρίζομαι ένα ε, πρόγραμμα 7 δις ευρώ που βεβαίως εντάσσεται στα μεγάλα, προβλήματα και, μεγάλα προγράμματα και φοβούμαι ότι θα αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους προγράμματα. Τέτοιου είδους προβλήματα, συγγνώμη, με τα μεγάλα προγράμματα. Στόχος θα πρέπει να είναι η τροποποίηση της αρχιτεκτονικής ε, για την ε, προγραμματική περίοδο 2007-2013, αλλά όπως ε, έλεγα και οι προηγούμενοι ομιλητές, οι τροποποιήσεις σε, οι τροποποιήσεις ε, μπορεί να έχουν ε, ε, ικανοποιητικό θετικό αντίκτυπο προς το τέλος της προγραμματικής περίοδου. Εμείς έχουμε και κάποιες προτάσεις. Πρώτα απ' όλα η αξιοποίηση των όσων γίνονται ή θα γίνουν στην προγραμματικη περιοδο περίοδο 7-13. Ε, οι επιθεωρήσεις ε, θα πρέπει να ε, αφορούν συγκεκριμένη προστεθέμενη αξία θα πρέπει οπωσδήποτε να μειωθεί η ανάγκη για μείωση του κόστους επί των δικαιούχων δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε επιπλέον επιβαρύνσεις και επιπλέον γραφειοκρατικά αχθη. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω ότι η παρουσίασή μου θα βρίσκεται στη διάθεση οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να τη διαβάσει εν και επίσης να πω τελειώνοντας ότι εάν θέλουμε να ξεπεράσουμε την παρούσα κρίση η οποία σφίγγει και συνθλίβει την ε, Ευρωπαϊκή Ήπειρο, θα πρέπει βεβαίως να σεβαστούμε τους κανόνες. Όταν όμως οι κανόνες πληθαίνουν, τότε οι εδαφικές ε, οντότητες κινδυνεύουν να πάνε από το κακό στο χειρότερο. Η πρόεδρος είπε ότι είμαι και υπεύθυνο ε, του γραφείου της ε, καμπάνιας στην Ευρωπαϊκή, στις Βρυξέλλες. Ο ε, Μονέ έλεγε ότι οι άνθρωποι γίνονται καλύτεροι όταν το πλαίσιο στο οποίο κινούνται είναι καλύτερο. Να Και το λέω για να θυμηθούμε λίγο και τους ε, πατέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον έτσι ώστε και οι περιφέρειες να βελτιωθούν όσο γίνεται περισσότερο στα πλαίσια της βελτίωσης των ταμείων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα προχωρούμε στον επόμενο μιλητή από τη Βουλγαρία, τον κύριο Μπέριν Μόλοφ, από τη Βέλγερ Κονσάλτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, για μένα αποτελεί τιμή ε, όσο και μεγάλη ευθύνη η ευκαιρία που έχω να συμμετέχω εδώ στην ακρόαση αυτή για την επόμενη προγραμματική περίοδο μετά το 2013 και το μέλλον της ε, πολιτικής συνοχής. Εγώ θα περιοριστώ στην ε, εμπειρία μου που έχω σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικού σχεδιασμού. Στόχο έχουμε να εφαρμόζουμε σωστά προγράμματα, καλά σχεδιασμένα για να έχουμε ε, αποτελέσματα αηφόρα και βιώσιμα προς το δημόσιο συμφέρον. Έχω κάνει μια σειρά διαφανειών, ελπίζω να τις δούμε. Εγώ είμαι αρχιτέκτονας, έχω σπουδάσει, αλλά κατά τη διάρκεια της ε, σταδιοδρομίας μου βασικά ε, στράφηκα στην πολεοδομία στρατηγικές προγράμματα, σχέδια, έργα ε, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στη χωροταξία, ε, σε τοπικό επίπεδο και περιφερειακό επίπεδο, ε, βιώσιμη και αηφόρο ανάπτυξη των πόλεων και εφαρμογή των πολιτικών συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τελευταία δύο χρόνια συμμετείχα στην εκπόνηση της βουλγαρικής θέσης για τη στρατηγική του Δουνάβεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρω τη στρατηγική αυτή του Δουνάβεως διότι θεωρώ ότι η μεθοδολογική προσέγγιση στην κατάρτιση ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα στάδιο και μια φάση για το νέο νομοθετικό πακέτο το οποίο σήμερα μας απασχολεί. Θα ήθελα να κάνω ε, σχόλια σε δύο σημαντικές ε, ενότητες. Αηφόρος αστική ανάπτυξη μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού και τοπική ανάπτυξη με βάση τοπικές κοινότητες ε, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε ειδικέ περιοχές. Πιστεύουμε ότι οι προτάσεις για τη μελλοντική πολιτική συνοχής είναι μια καλή αφιτηρία για να εφαρμόσουμε μια φιλόδοξη πρόταση για ένα πρόγραμμα αστικής ανάπτυξης. Μπορεί να είναι μια μεγάλη κινητήρια δύναμη που θα είναι τελικά προς όφελος όχι μόνο του αστικού πληθυσμού στα μεγάλα κέντρα, αλλά ε, όλου του πληθυσμού ενός κράτους. Γι' αυτό καλωσορίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ειδικά προγράμματα για τις αστικές περιοχές που θα επικεντρώσουν τη χρηματοδότηση σε μια στρατηγική για χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, βιώσιμες ε, αστικές συγκοινωνίες, βελτιώσεις για το αστικό περιβάλλον και οικονομική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών. Βεβαίως, εδώ χρειάζεται μια κάποια ευελιξία ε, στην εφαρμογή της θεματικής συγκέντρωσης. Βλέπετε στη διαφάνεια αυτή τις μεγάλες βουλγαρικές πόλεις που είναι μεγάλα αστικά κέντρα. με ολοκληρωμένα προγράμματα αναδόμησης, ανοικοδόμησης και αναζωγόνησης των πόλεων. Διάφορα έργα που θα ε, χρηματοδοτηθούν από τα, το ΕΣΠΑ της Βουλγαρίας για το επόμενο διάστημα, την επόμενη προγραμματική περίοδο. Ανακοδόμηση λοιπόν και ανάπτυξη των πόλεων. Αυτό είναι καινοτομία ε, στη βουλγαρική πραγματικότητα και στον τρόπο με τον οποίο εργάζονται και συνεργάζονται οι διάφοροι φορείς. Θεωρούμε αυτό το πρόγραμμα ως ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο στο χώρο και στο χρόνο ε, με συνοχή και συνεργασία διαφόρων τομέων. Έχουμε μια σειρά συμμετεχόντων ε, που από κοινού ε, ακολουθούν ένα κοινό στόχο. Με όραμα, με στρατηγική για την αστική ανάπτυξη και ιδιαίτερα ε, σε συγκεκριμένες προτεραιότητες. Για μας η ιδιαιτερότητα της ολοκληρωμένης προσέγγισης και του ολοκληρωμένου σχεδιασμού ποια είναι. Περιλαμβάνει όχι μόνο σχέδια χωροταξίας, πολεοδομίας και επενδύσεων, αλλά διάφορους ε, φορείς που συμμετέχουν, διάφορες οργανώσεις οικονομικές, κοινωνικές που ε, συνεισφέρουν στη γενική αηφορία και εξασφαλίζουν την προστιθέμενη αξία. Στη Βουλγαρία η ανάπτυξη ε, και το πρόγραμμα αυτό για την ανοικοδόμηση και ανασυγκρότηση των πόλεων συνδέεται με το λειτουργικό επιχειρησιακό πρόγραμμα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, αλλά και άλλα ε, προγράμματα για τις πόλεις. Εκτός από τα κονδύλια που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ολοκληρωμένα σχέδια θα χρησιμοποιήσουν και άλλες δυνατές πηγές χρηματοδότησης και μηχανισμούς, όπως είναι η προσέλκυση ιδιωτικού κεφαλαίου και οι ΣΔΙΤ, ε, συμπράξεις ε, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Σας δείχνω εδώ σε αυτή τη διαφάνεια πώς εντάσσεται αυτό το ολοκληρωμένο σχέδιο στον εθνικό μας σχεδιασμό. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για το δυναμικό που υποστηρίζεται από αυτό που είναι γνωστό ως ε, ολοκληρωμένη δαφική επένδυση, το ITI. Αυτό είναι ένα νέο μέσο και μια νέα πρωτοβουλία που θεωρεί την εδαφική επένδυση ως ένα νέο μέσο σε διάφορα προγράμματα και με την επένδυση αυτή μπορούν να συνδυαστούν κονδύλια από διάφορες πηγές. Έχουμε διάφορες λειτουργικές αστικές περιοχές ε, αρχής γενομένης από τη γειτονιά, από τη συνοικία μέχρι και ευρύτερα αστικά κέντρα, πολλές φορές μπορεί να είναι και παρακείμενες πόλεις ή υπαίθριες περιοχές. Προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τουλάχιστον το 5% των κονδυλίων για κάθε κράτος μέλος ε, από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το ΦΕΝΤΕΡ, να πηγαίνει στην αστική ανάπτυξη. μέσω της ε, ολοκληρωμένης εδαφικής επένδυσης. ITI. Η διαχείριση ανατίθεται πλέον στις πόλεις και αυτό είναι μεγάλη πρόκληση και χρειάζεται προσπάθεια για να οικοδομηθεί η ικανότητα καν διαχείρισης που είναι απαραίτητη. Το είπαν και οι προλαλήσαντες αυτό. Επιτρέψτε μου να σας πω ε, δύο λόγια τώρα για κάτι πολύ σημαντικό ως εξέλιξη στη Βουλγαρία που είναι η προετοιμασία συμμετοχής, αυτό που είναι γνωστό ως ε, η τοπική ανάπτυξη που βασίζεται στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό μπορεί να είναι πραγματικά η βάση για μια υφόρο ανάπτυξη. Τι σημαίνει αυτό. σε μια επικράτεια, σε ένα έδαφος και περιφέρεια με ειδικά χαρακτηριστικά να λαμβάνει ο τοπικό πληθυσμό ή οτά οι ομάδε δράση, την ανάπτυξή του. Αυτοί μπορεί να είναι εκπρόσωποι του δημοσίου τομέα, του ιδιωτικού, μη κυβερνητικών οργανώσεων και ε, σε επίπεδο λήψης αποφάσεων και γενικότερα. Και σε αυτά τα συμβούλια, καμία από τις ομάδες αυτές δεν έχει περισσότερο από 49% δικαιώματα ψήφου. Προσπαθώ λοιπόν εδώ να σας δείξω ομάδες κοινοτήτων τέτοιες που έχουν κοινά σχέδια για να αναπτύξουν ε, μια πρόταση ε, εντός ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος για αναπτυξιακά σχέδια. Έτσι, επιλέγονται και χρηματοδοτούνται έργα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που θα έχουν με αυτόν τον τρόπο πολύ μεγαλύτερη απόδοση από ό,τι συμβαίνει σήμερα. Η επόμενη διαφάνεια, ελπίζω να ε, τη βλέπετε όλοι, μας δείχνει και προσπάθησα να περιγράψω τη δυνατότητα που έχουν τα διάφορα ταμεία να χρηματοδοτούν στρατηγικές με συνεργασία των ενδιαφερομένων φορέων. Και ειδικά έργα και project σε διάφορους τομείς πολιτικής συνοχής και σε διάφορες περιοχές. Επειδή όμως τελειώνει ο χρόνος μου, θα ήθελα να σας δείξω ένα νέο παράδειγμα της περασμένης εβδομάδας μάλιστα, τι έγινε στη Βουλγαρία, στη Νότια Βουλγαρία. Είναι μια διασυνοριακή περιφέρεια, παραμεθόριος. Ε, με 8 κοινότητες ε, είναι ε, στην κοιλάδα του ποταμού Μέστα, του ποταμού Νέστου, στα ελληνικά. Ε, λοιπόν, εκεί συνεργάζονται 8 κοινότητες για να προετοιμάσουν ε, την ε, πρόταση για την άτυπη λεγόμενη περιφέρεια. Συνεργάζονται όλοι οι ενεχόμενοι, οι ενδιαφερόμενοι φορείς και θα προετοιμάσουν μια στρατηγική για αστική ανάπτυξη για την επόμενη προγραμματική περίοδο και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Μόλοφ για τα σχόλιά σας σχετικά για τη διαχείριση και τώρα θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Λοχάιντε. Ε, κύριε καθηγητά, ελπίζω ότι πρόφερα σωστά το όνομά σας γερμανικά και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ. Έχουμε προετοιμάσει μία μικρή παρουσίαση την οποία θα ξεκινήσουμε ε, σχετικά με την υποδομή ε, της ε, τραπέζης της ΕΣΥΣ η οποία προωθεί και την γεωργία και την περιφέρεια του κρατηδίου και ξεκινώ με τα βασικότερα κοινά προγράμματα, δηλαδή απλοποίηση της ε, πολιτικής συνοχής, ερεσιμότης ε, και ε, προώθηση. Αυτά ήταν οι επιταγές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ στην απλοποίηση και την αποδοτικότητα και να εξετάσω και το θέμα των ε, μέσων ε, ε, χρηματοδοτήσεως. Υπάρχουν και συμμετέχοντες που μου απίφθηναν το λόγο και που ασχολούνται με παρεμφερή προβλήματα, οπότε θα συνεχίσω εκεί που σταμάτησαν. Η συνοχή πρέπει να φροντίσει ώστε έως το, την 31 Δεκεμβρίου του 2021 όλες οι ανταλλαγές απόψεων να γίνονται και πληροφοριών να γίνονται ε, ψηφιακά μέσω του διαδικτύου, πράγμα το οποίο θα βελτιώσει την ε, ε, απόδοση και ιδίως όσον αφορά τις, τα στοιχεία της, των εποπτικών αρχών, αλλά θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που δημιουργεί αυτό το σύστημα και αυτό διότι κατερχόν ε, δεν μπορούμε να σεβαστούμε πιστεύω την προθεσμία μέχρι τέλους του 2014 ε, είναι μικρά τα γράμματα και νομίζω ότι δεν ε, θα μπορέσετε να το διαβάσετε αλλά ε, διότι χρειάζεται ένα τόσο περίπλοκο πρόγραμμα ηλεκτρονικό ώστε να χρειάζεται τουλάχιστον 36 μήνες από όταν θα γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν χαιρετίζουμε την πρόταση της Δανικής Προεδρίας και την πρόταση να μετατεθεί η προθεσμία μέχρι το τέλος του 2016 αλλά εμείς πιστεύουμε ότι ουσιαστικά για να είμαστε ρεαλιστές χρειαζόμαστε περιθώριο μέχρι το 2017 για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας διότι θα υπάρχουν και οι κατεξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες θα χρειαστεί να καταρτιστούν αφού ληφθούν οι αποφάσεις. Επιπλέον υπάρχει και το θέμα των ε, πόρων ε, και χρηματοοικονομικών και σε ανθρώπινο δυναμικό. Η χρηματοδότηση ενός ε, τόσο εκτενούς προγράμματος είναι δύσκολη και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στηρίξει ε, με τεχνική βροήθεια το πρόγραμμα. Για να σας δώσω κάποια ιδέα, ε, είχαμε ζητήσει ε, επιδόμα την προηγούμενη φορά 750.000 ευρώ συγκεκριμένα αλλά εάν προσαρμόσουμε το πρόγραμμα αυτό ε, θα χρειαστεί ε, να προσαρμόσουμε οι 28 μέτρα, δηλαδή μιλάμε για εξαψήφιους αν όχι εφταψήφιους αριθμούς και άρα θα πρέπει να πούμε ότι ε, όποιος επιθυμεί κάτι τέτοιο θέλει να δει, θέλει να μας πει πώς θα, χρηματο, θα χρηματοδοτηθεί ε, και όποιος το παραγγέλνει θα πρέπει να μπορεί να το πληρώσει. Και τα τεχνικά αυτά θέματα προς το παρόν δεν τα έχουμε λύσει. Όσον αφορά την απλοποίηση. Έχω πολλά παραδείγματα αλλά θα τα παρακάμψω τώρα για να μπορέσω να κερδίσω το χαμένο χρόνο. Αλλά αναφέρομαι στην πιστοποίηση. Διότι για τον ε, έλεγχο και την διαχείριση των προγραμμάτων χρειάζεται μία αρχή η οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη στα Υπουργεία και θα υπάρχει και πάνω από αυτήν μία αρχή πιστοποιήσεως που θα πιστοποιεί αυτή την υπηρεσία. Επιπλέον λοιπόν ε, θα χρειαστεί να υπάρχει μία υπηρεσία στο Υπουργείο που θα εφαρμόζει τα διαρθρωτικά μέτρα και θα χρειαστεί χρηματοδότηση, πράγμα το οποίο οδηγεί σε μία επιπρόσθετη διοικητική δαπάνη, χωρίς όμως από εκεί να υπάρξει κάποιο όφελος. Άρα όλες αυτές οι ελεγκτικές και εποπτικές αρχές κατά τη γνώμη μας δεν είναι, ε, δεν είναι πολύ αποδοτικές και θα πρέπει να βελτιωθούν ποιοτικά. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει πρόθεση της γεωργίας μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και θα ήθελα να ρωτήσω, εκεί υπάρχουν τόσο πολλά περισσότερα ασφάλματα ώστε να δικαιολογούνται τόσο περισσότερες θέσεις. Θα πρέπει επιπλέον να είναι επικοδομητικά διότι δεν προσπαθούμε να απλοποιήσουμε απλώς τις ρυθμίσεις αλλά και να τις αντιμετωπίσουμε με ένα ενημαίο τρόπο. Επίσης όλα αυτά ελέγχονται από το Γερμανικό Ελεγκτικό Συνέδριο, από το Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΣΥΣ από την ε, ε, υπηρεσία υπάρχουν δηλαδή πολλαπλοί έλεγχοι και αναρωτιέμαι είναι αναγκαίοι όλοι αυτοί ή μπορούν να συνοψιστούν και να περιοριστούν. Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα με τις προτάσεις ε, ε, του κανονισμού έχουν, ε, ε, ε, έχουν δημιουργηθεί οι χρηματοδοτικές προτάσεις και χαιρετίζουμε το μέτρο αυτό διότι όντως υπάρχει μία απλοποίηση, είναι πολύ πιο εύκολο να τα διεκπεριώσουμε. Υπάρχει το προσόν των μέσων που μπορούν να αποπληρωθούν, μπορεί να υπάρχει μόχλευση με ε, ιδιωτικά κεφάλαια και να αυξηθεί η αποδοτικότητα και μειώνοντας και τα λάθη και ε, έχοντας μία πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση. Επιπλέον πρέπει να αποφύγουμε τις τρευλώσεις της αγοράς. Αυτή είναι μια σαφής βελτίωση την οποία διαπιστώνουμε, αλλά πρέπει να πούμε ότι όσον αφορά την εφαρμογή, μέχρι στιγμής στις προτάσεις βλέπουμε ότι υπάρχει άνηση αντιμετώπιση των εναλλακτικών λύσεων χρηματοδοτήσεως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα συνδέει με σημαντικά κίνητρα για να μπορέσει να τα εφαρμόσει. Αυτά δεν μου φαίνονται πλήρως ε, ρεαλιστικά και δεν αντιλαμβάνομαι γιατί υπάρχει αυτή η ε, ασυνέπεια. Θα μπορούσαν να ισχύσουν όλα αυτά και να εφαρμοστούν πολύ πιο ε, ικανοποιητικά και πιστεύω ότι η τα θεσμικά όργανα τα οποία εφαρμόζουν τις διατάξεις γνωρίζουν τις ανάγκες και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα χρηματοδοτικό μείγμα που θα προσαρμόζεται στις ανάγκες των χρηστών και να χρησιμοποιήσουν και ιδιωτικά κεφάλαια για την συμπλήρωση των ε, ταμιακών φόρων. Ε, προσπαθώ τώρα να συνοψίσω. Σας ανέφερα διάφορα παραδείγματα και αναρωτιέμαι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέτυχε το στόχο της. Ουσιαστικά νομίζω ότι η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εναρμονίσει ε, τα, ε, τις χρηματοδοτήσεις αυτής βαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Η εναρμόνιση της ρυθμίσεως των ταμείων θα απλοποιήσει την εφαρμογή θα μπορέσει να επιτρέψει να υπάρχουν ενιαία προγράμματα για την αναφορά, για τη διεκπαιρέωση, να μειώσει το κόστος της διαθέσεως της χρηματοδοτήσεως. Δηλαδή θα υπάρξει όντως απλοποίηση αλλά δεν αρκεί. Και τα παραδείγματα τα οποία ανέφερα για την περιοχή μας δείχνει ότι θα πρέπει να είμαστε πιο απλοί και όχι το αντίστροφο παραδείγματος χωρίν μέχρι στιγμής είδαμε ότι ε, επιτύχαμε και χωρίς ε, τα μέτρα αυτά. Η νέα κατεύθυνση θα δημιουργήσει και νέες απαιτήσει. και μειώνουμε με ε, τα ελεγκτικά μέτρα όχι όμως επαρκώς και χρειάζεται μεγαλύτερη αποθηκευτική ικανότητα και αυτό που είπε ο κύριος Μέντες ε, ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση με τη δική μας ε, και αν ε, αναφερθώ σε αυτά που είπε ο κύριος Τρίλινγκ για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μπορώ να προσθέσω ότι αν υλοποιήσουμε το στόχο αυτό θα πρέπει συγχρόνως να εξασφαλίσουμε ότι στην πρακτική θα συγκεντρωθούν τα, οι πόροι σε λιγότερους στόχους για να μπορέσουμε να τους επιτύχουμε διότι θα χρειαστούν ε, μαζική ε, χρηματοδότηση ε, διότι αν έχετε 50 μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή 50 κοινοτικές επιχειρήσεις δεν θα μπορέσετε να τις προωθήσετε όλες με τον ίδιο τρόπο. Θα πρέπει να προωθήσουμε με μονομένους πιο σημαντικούς στόχους και όχι όλους μαζί και Τέλος θα πρέπει να υπάρχει ενιαία ερμηνεία ε, και να υπάρχει ε, ασφάλιση ασφάλεια προγραμματισμού. Πράγμα το οποίο έχουμε δει και στο παρελθόν. Αν υπάρχουν εκ των υστέρων τροποποιήσεις, αυτό είναι όντως πολύ βραβερό και χρειαζόμαστε ε, συγχρόνως συμμετοχή του Κοινοβουλίου και διαφάνεια κατά τρόπον ώστε να μην υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις γιατί όταν υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις εάν οι εφαρμοστικές διατάξεις ε, δεν είναι απλές δεν θα επιτύχουν το στόχο για τον οποίο εκπονήθηκαν. Γι' αυτό και πρέπει να δούμε πώς ε, θα διατυπωθούν οι ε, εφαρμοστικές διατάξεις. Έχουμε και άλλα ε, σχόλια. Θα σας στείλουμε ένα έγγραφο μέσω της γραμματείας όπου σχολιάζουμε πιο, σε πιο πολλές λεπτομέρειες ορισμένα θέματα και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Λοχάιντε και για την επικριτική σας ανάλυση και εξέταση της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα παρακαλέσω τώρα την Κομισιόν να λάβει θέση, εάν παρευρίσκεται, ποιος θέλει να αναλάβει αυτό το έργο. Αποουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, όχι, ο κύριος Μάρτιν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, για την ευκαιρία που μου δίνετε Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη η σειρά και πλούσια των παρεμβάσεων και είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς. Και ξέρω ότι δεν έχουμε και πολύ χρόνο γιατί θέλετε να το συζητήσετε. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στα βασικά σημεία όπως τα βλέπω εγώ. Αυτό που είπε πρώτος ο δόκτωρ Ζούλεκ για αλλαγή υποδείγματος και τρόπου προσέγγισης στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στρατηγική διεύθυνση του προγραμματισμού. Και απάντησε αρνητικά εγώ θα τόνιζα το εξή, χωρίς να χρησιμοποιήσω την ίδια ορολογία. Αν θέλετε να το πω πιο απλά, με πιο απλά λόγια, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι προτάσεις μάλιστα περιλαμβάνουν θεμελιώδη αλλαγή στην προσέγγιση, ε, στο στρατηγικό προγραμματισμό και στην ε, χάραξη και εκτέλεση πολιτικής συνοχής συνδέεται με τις προτεραιότητες το 2020 και με τις επιδόσεις και με τα αποτελέσματα. Έχουμε μια σειρά από μηχανισμούς τώρα στην προτάση μας που αν ε, ευδοκιμήσουν θα αποτελέσουν πραγματικά καμπή στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η πολιτική συνοχής. Είναι μια νέα λογική στην επέμβαση και στις παρεμβάσεις. Δηλαδή θα ε, είμαστε πάρα πολύ στοχευμένοι με συγκεκριμένους στόχους. Και στόχοι τι είναι. Δεν είναι να γράφουμε συγκεκριμένες λέξεις για την αποστολή των ταμείων στον κανονισμό, αλλά να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό που θα εξασφαλίζει ότι θα χρησιμοποιούνται με ένα συγκεκριμένο τρόπο τα κονδύλια, με σωστά σχεδιασμένα επιχειρησιακά προγράμματα και τα κονδύλια θα συνδέονται με σαφώς καθορισμένους στόχους. Γι' αυτό μιλούμε για θεματικές ενότητες και θεματικούς στόχους για το 2020 και έχουμε φτιάξει το πρόγραμμα έτσι ώστε οι υπεύθυνοι να εντοπίζουν και να ταυτοποιούν τους στόχους για κάθε άξονα προτεραιότητα στο πρόγραμμα και να συνδέονται έτσι λοιπόν και οι δείκτες αποτελεσμάτων με αυτούς τους στόχους. Υπάρχει ένας μηχανισμός ακριβώς για να ταυτοποιούνται τα αποτελέσματα, οι στόχοι και να παρακολουθείτε και να ελέγχετε αυτή η διαδικασία κατά πόσο έχει επιτευχθεί. Οι δείκτες είναι πολλοί. Είναι ένα ολόκληρο σύνολο Το ανέφερε ο κύριος Τρίλινγκ. Αλλά είναι σημαντικό να δούμε τη συνολική δέσμη. Πώς χτίζεται ένα πρόγραμμα, οι προτεραιότητες από τους ειδικού στόχους μέχρι τα αποτελέσματα και τους δείκτες που έχουν ταυτοποιηθεί και επίσης τους στόχους του, του, του τελικού προϊόντος, το output, για να δούμε πώς οι μεμονωμένες δράσεις υλοποιούνται και πού καταλήγουν, τι παράγουν και ποια αποτελέσματα. Η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής δεν είναι χρήσιμο ούτε σκόπιμο εκ των προτέρων να έχουμε στόχους ως προς το αποτέλεσμα. Θα πρέπει αυτά να τα εντοπίζουν εκείνοι που θα σχεδιάσουν το πρόγραμμα και να τα συζητούν και να τα διαπραγματεύονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό θα είναι πραγματικά σημαντικό τμήμα της όλης διαπραγματευτικής διαδικασίας. Και αυτό συνεχίζεται με το λεγόμενο πλαίσιο επιδόσεων. Δηλαδή εκεί θα ε, συλλαμβάνονται κατά κάποιο τρόπο οι δείκτες αποτελέσματος και θα υπάρχει ένας μηχανισμός που θα εξασφαλίζει τις επιδόσεις. Αυτό θέλουμε. Είναι γεγονός και έχετε δίκιο ότι υπάρχουν δυσκολίες. Και σωστά είπε ο Δόκτωρ Ζούλεκ ότι ορισμένα πράγματα είναι προβληματικά και πρόκληση όντως. Το ξέρει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά το, επειδή υπάρχουν προβλήματα λοιπόν και ενδεχομένως δυσκολίες δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και να μην επιζητούμε ακριβώς ε, την επίτευξη αυτού του μηχανισμού για να αλλάξει η εστίαση. Όχι απλώς να απορροφούμε κονδύλια, αλλά να φτάνουμε σε πραγματικούς στόχους που τους έχουμε εντοπίσει εκ των προτέρων. Και αυτό θα γίνει ακριβώς με τους βασικούς δείκτες και δείκτες αποτελέσματος, output ή ε, ε, result indicators είναι και ένα ζήτημα χρόνου. Αν θέλει κανείς να αναθεωρεί τη διαδικασία για να κάνει κάποιες αλλαγέ. δεν θα πρέπει να περιμένει το τελικό αποτέλεσμα ε, το τέλος προγραμματική περίοδου, αλλά και το ενδιάμεσο προϊόν. Αλλάζουμε βεβαίως κατεύθυνση και είναι σαφής αυτή η αλλαγή. Και κατά την άποψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό είναι πραγματικά θεμελιώδες ως αλλαγή στην προσέγγιση. Τώρα, για το θέμα της απλοποίησης. Και αυτό είναι βασικό θέμα της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν και άλλες δημοσιεύσεις που ορίζουν ρητός ε, τι εστί απλοποίηση. Για τους δικαιούχους και ε, για το θέμα της ηλεκτρονικής συνοχής. Σε ό,τι αφορά την απλοποίηση για τις διαχειριστικές υπηρεσίες, ποιο είναι η δοκιμή, το τεστ. Εάν αυτό που ζητεί ο κανονισμός είναι δικαιολογημένο. Υπάρχουν και όρια στην απλοποίηση μιας διαχείρισης ε, και ενός management, αν θέλει κανείς να εξασφαλίζει ότι δαπανώνται σωστά τα κονδύλια. Εξού και η ρεσιμότητα και το πλαίσιο επίδοση. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το κόστος του να μην το κάνουμε αυτό, ότι κάθε ευρώ πιάνει τόπο. Είναι πολύ μεγαλύτερο και αν θα πρέπει να σταθμίσουμε αυτά τα πράγματα, να δούμε ε, ποια είναι η κατάσταση. Για την ηλεκτρονική συνοχή Νομίζουμε ότι τώρα με την ψηφιακή ατζέντα και τους στόχους της αυτό ευθυγραμμίζεται. Πολλά κράτη-μέλη έχουν μπει εκεί, υπάρχει χρηματοδότηση από την παρούσα προγραμματική περίοδο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πρόθυμη να δώσει και τεχνικές συμβουλές για αυτό το θέμα. Τέλος, για το σύστημα Ε, κοινοποίησης για να δείξουμε ότι πραγματικά προχωρούμε προς την κατεύθυνση αυτή και φεύγουμε και καταλείπουμε τις δυσκολίες που έχουμε κάθε χρόνο για τα επίπεδα σφάλματος, δεν μπορούμε να σταματήσουμε εκεί σε μια αποτελμάτωση. Χρειάζεται βασική αναδιάρθρωση, βέβαια με μεγάλη συνέχεια στη βασική αρχιτεκτονική. Έχουμε όπου αυτό γίνεται streamlining ας πούμε, τις αιτήσεις εκθέσεις εφαρμογής, αλλά τα στοιχεία της πιστοποίησης ακριβώς ενισχύουν τους ελέγχους εκ των προτέρων και τα κράτη-μέλη είναι σαφώς υπεύθυνα για τους φορείς που έχουν οριστεί και για να τους ελέγχουν. Και οι οι λογαριασμοί είναι κάτι το φυσιολογικό για όλους τους οργανισμούς. Κάθε οργανισμός έχει αιτήσιους λογαριασμούς. Ε, αυτό είναι σημείο αναφοράς για τις δηλώσεις και τις διασφαλίσεις που δίνονται. Η διαχείριση των προγραμμάτων μπορεί να γίνει έτσι. Για να ενισχυθεί. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ja, herzlichen Dank. Ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα να ακούσουμε τώρα τις αντιδράσεις στην ε, ε, παρουσίαση, στις παρουσιάσεις των εμπειρογνωμόνων και σας δίνω τώρα το λόγο σε εσά σαν ευρωβουλευτές. Μέχρι στιγμής έχουμε δύο που ζητούσαν το λόγο. Παρακαλώ όλους να μην κάνουν ομιλίες αλλά να πρόκειται για ερωτήσεις. Ο πρώτος υποψήφιος είναι ο Γιάνν Όλμπριχτ, ε, ο οποίος είναι ένας από τους λίγους ο οποίος γνωρίζει όλο το σύνολο αυτό που είναι τόσο περίπλοκο σαν εμπειρογνώμων. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια κύριε Πρόεδρε. Ένα ερώτημα. Το πρώτο μου ερώτημα απευθύνεται στον καθηγητή Τζον Μάκνορ. Δηλαδή, ε, είπατε ότι το CFF δεν έπρεπε να έχει ε, να μην είναι πράξη κατά εξουσιοδότηση και τώρα όμως έχει γίνει. Ε, τι πιστεύετε, πιστεύουμε ότι το κείμενο το οποίο έχουμε για το CSF ε, είναι μία κατεξουσιοδότηση ε, πράξη, δηλαδή το Common Strategic Framework, το κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Άρα ποια είναι η σημερινή σας αντίδραση. Πιστεύετε ότι πρέπει να παραμείνει πρωτογενής νομοθεσία. Δεύτερον, στον κύριο Μάρκου Στρίλινγκ σχετικά με τους δείκτες. Από ό,τι κατάλαβα ε, και δεν ξέρω αν κατάλαβα σωστά, εσείς θεωρείτε ότι οι δείκτες είναι ισότιμοι με τους θεματικούς στόχους. Οπότε αυτό μου φαίνεται λογικό και αυτό το οποίο έχουμε εις το πλαίσιο, στο περιφερειακό πλαίσιο αναπτύσσεως θα πρέπει επίσης να ισχύσει. Ε, μπορούμε να συμβιβάσουμε τις προτεραιότητες με τους δίκτες, διότι κατά τη γνώμη μου διαφορετικά χαθήκαμε. Θα μπερδευτούμε. Εάν λοιπόν ε, διαγράψει κανείς όλους τους δείχτες από το πλαίσιο, ε, το περιφερειακό πλαίσιο ανάπτυξης ε, τι θα γίνει. Εγώ είμαι υπέρ της διαγραφής από αυτό το πλαίσιο. Αλλά εσείς λέτε να ενσωματώσουμε τους δείχτες στο γενικό κεφάλαιο. Επίσης, ε, ε, ένας άλλος ομιλητής είπε ότι οι παρατηρήσεις του βασίζονται στις ε, νέες προτάσεις του δημοσιονομικού κανονισμού. Ενώ βλέπουμε ότι η διεργασία αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Πιστεύετε λοιπόν ότι αυτή η προετοιμασία θα εμποδίσει το σύνολο γιατί πιστεύουμε ότι ε, υπάρχει μία, ένα στοιχείο μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Εσείς κάπως τα έχετε μπερδέψει και τα καθιστάτε πιο περίπλοκα. Αντιλαμβάνομαι ότι έχετε προεξοφλήσει ορισμένες ε, επιπτώσεις. Σωστά κατάλαβα. Ευχαριστώ. Εντάξει, Κατά σειράν των ετούντων θα ακούσουμε ακόμη δύο μιλητές και στη συνέχεια θα δώσουμε το λόγο στους εμπειρογνώμονες. Ε, καταρχήν έχουμε τον κύριο Βανίσεροι και μετά την κυρία Κρέλ. Ευχαριστώ πολύ. Και όλα τα σχόλια τα οποία κάνουμε συνήθως. Λοιπόν, Βλέπω τη σελίδα 6 του εγγράφου που σας έδειξα και εδώ ε, αναφέρεται η σαφής ανάγκη σε όλου του πλαισίου. Εσείς ο εμπειρογνώμονας έχετε παρακολουθήσει χρόνια τον τρόπο με τον οποίο εμείς ε, ε, υλοποιούμε και την στρατηγική μας ε, να προχωρήσει, μπορεί να προχωρήσει πάντως με τον τρόπο τον οποίο είναι διατυπωμένη τώρα. Εσείς λέτε ότι θα πρέπει ε, να απλουστευθεί. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη, υπάρχει αποσαφήνιση. Η Κομισιόν έρχεται με νέες ε, προτάσεις διαρκώς. Πόσο βαθιά είναι τα προβλήματα τα οποία αναφέρεται στη σελίδα 6. Έπειτα, σε μια περίοδο κρίσης. Ε, πιστεύουμε ότι αυτή η συγχρηματοδότηση ότι θα οδηγήσει τελικά σε κάποια, δηλαδή θα, θα βρεθούν κάποια ε, δημόσια χρήματα, κάποια εθνικά χρήματα έτσι ώστε να βελτιωθεί πραγματικά ε, η ζωή των πολιτών που ζουν στις πόλεις ή τέλος πάντων στις περιοχές γιατί διαφορετικά θα χρησιμοποιηθούν λιγότερο τα ταμεία, οι πόροι δηλαδή των ταμείων. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό. Και μία ερώτηση στον συνάδελφο από την, τον εκπρόσωπο μάλλον της ε, ε καμπανίας. Είχαμε, είχαμε τον Υπουργό Μπάρκα, ο οποίος ε, είπε ότι δημιουργήθηκε στην Ιταλία μια νέα δυνατότητα, έγιναν ρήξεις και τελικά παίρνοντας ας πούμε κάποια χρήματα από τις ε, μεταφορές και μετά χρησιμοποιώντας τα χρήματα αυτά μαζί με εθνικούς πόρους ε, λειτουργήσαν καλύτερα τα συστήματα. Ακούσαμε ότι είστε επικριτικός όσον αφορά τους, ε, τον νέο κανονισμό. Πιστεύω ότι για πρώτη φορά σε αυτήν την εταιρική σχέση ε, θα είναι άμεσα εμπλεκόμενο και το κράτος. Τέλος, ο κύριος Τέλινγκ μας μίλησε για δείκτες και για δείκτες αποτελέσματος τι, ποια είναι η άποψή σας όσον αφορά την ίδια την επίδοση. Κωνσταντσα Κρέλ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες, ενδιαφέρουσες οι παρεμβάσεις. Επίσης αντανακλούν και αυτά που συζητούμε εμείς στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μας εδώ και μήνες ήδη. Δεν θέλω να επαναλάβω τίποτα που ρώτησαν οι προλαλήσαντες. Εμένα με απασχολεί πάντα πάρα πολύ και με ενδιαφέρει το θέμα της απλοποίησης. Θαυμάσια ακούγονται όλα αυτά. Να, αν ελέγχουμε 5-6 φορές το ίδιο σχέδιο, το ίδιο έργο, γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αμοιβαία, αμοιβαία συγγνώμη, ε, κάτι που έχει ελέγξει κάποιος άλλος. Πού θα το γράψουμε όμως, δεν μπορούμε αυτό να το γράψουμε στον κανονισμό, ότι το εκάστοτε ελεγκτικό συνέδριο του Ομόσπονδου Κρατηδίου ή το κράτους ή το ε, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο το έχει ελέγξει, θα πρέπει αμοιβαία να δέχονται τα πορίσματα του εκάστοτε ελεγκτικού συνεδρίου του τοπικού της κάθε χώρας. Δεν το καταλαβαίνω. Μπορεί να ακούγεται πολύ ωραίο, αλλά πώς θα το μεταφέρουμε και θα το εφαρμόσουμε στην πράξη στην πραγματικότητα. Εκεί έχετε πρόταση συγκεκριμένη. Λοιπόν, τώρα έχουμε τον πρώτο γύρο των απαντήσεων από τους εμπειρογνώμονες. Ποιος αρχίσει πρώτος, ο κύριος Πράτερ. Ich Παρακαλώ. σύντομες οι απαντήσεις, συντομότερες από τις ερωτήσεις, παρακαλώ. Θα το καταφέρουμε. Ναι, θα είναι ωραίες και σύντομες οι απαντήσεις. Στην πρώτη ερώτηση από τον κύριο Άλμπρεχτ. Έχοντας δει το πολιετές ε, πλαίσιο, ναι. Έχοντας δει το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, μπορώ να απαντήσω θετικά. Και το, αυτό το στρατηγικό πλαίσιο θα πρέπει να έχει, είναι ένα έγγραφο, κατά την άποψή μου, πιο, με μεγαλύτερη δύναμη και βλέπουμε ή, ήδη διαβλέπουμε πεδίο περαιτέρω ενδυνάμωσης σε διάφορα, ε, σε διάφορους τομείς. Χρειαζόμαστε δέσμευση, δεσμευτική δηλαδή η ηδη διαβλεπουμε πεδιο περαιτερω ενδυνάμωση σε διαφορα σε διαφορους τομεις χρειαζομαστε δεσμευση δεσμευτικη δηλαδη η σταση του ε, Συμβουλίου στο πλαίσιο αυτό. στα ερωτήματα που έθεσε ο κύριος Βανέστεροι, δεν είμαι σίγουρος εάν αναφερθήκατε στο ίδιο το στρατηγικό πλαίσιο ή ε, στον, ε, στο αποτέλεσμα παρατήρηση εκτός μικροφώνου στους στόχους, σε σχέση με τους στόχους ε, αυτά, θα συμφωνήσουμε με αυτά που είπε ο Νίκολας Μάρτιν. Υπήρξαν σημαντικές αλλαγές ε, σε σχέση με τα αναμενόμενα από την ε, πολιτική συνοχής και τα αποτελέσματα, ιδίως όσον αφορά τις περιφέρειες, χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια ένα από τα προβλήματα της ε, ε, πολιτικής συνοχής ήταν η, ο πολλαπλασιασμός των ε, στόχων και ο μη συντονισμός, η έλλειψη συντονισμού μεταξύ αυτών των πολιτικών. Ελπίζουμε λοιπόν και αναμένουμε, προσδοκούμε να υπάρχει καλύτερη ιεράρχηση όλων των στοιχείων σε σχέση με συγκεκριμένους στόχους ε, και ε, να δοθεί προτεραιότητα στους κατά προτεραιότητα στόχους ακριβώς. Δεν, ε, δεν ζητάμε απαραίτητα μία νέα πρόταση, ζητάμε σαφήνεια στην υφιστάμενη πρόταση. Είτε μέσω ενός νέου άρθρου, είτε μέσω της χρήσης υφισταμένου άρθρου για περαιτέρω αποσαφήνιση. Αυτό. Καλώς. Επόμενος επιρρογνώμων. Παρακαλώ, κύριος Γκαργίλη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου με το θέμα των ε, ε, στόχων ε, αποτελέσματος αλλά νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ευθυγραμμιστεί με την κρίση. Είναι δύσκολο να θέσει κανείς στόχους σήμερα ε, που ενδεχομένως σε δύο χρόνια δεν θα είναι, δύο-τρία χρόνια δεν θα είναι καθόλου οι ίδιοι. Ε, δεν αναφέρθηκα στο θέμα αυτό στην παρέμβασή μου, γιατί εκεί προσπάθησα να μιλήσω μονάχα για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα οι διαχειριστικές αρχές. Ο κ. Σόλμπρεχτ ακριβώς αναφέρθηκε στο μέλλον. Ναι, εμείς ακριβώς κάνουμε μια προβολή προς το μέλλον. Είναι περίεργο που το λέμε, αλλά έτσι είναι. Και οι οικονομικοί ελεκτές της ε, Επιτροπής ερμηνεύουν ήδη τις κανονιστικές προτάσεις ε, σαν να ήταν ε, ήδη κανονικός κανονισμός, ας πούμε. Και αναφέρθηκε σε αυτό και ένας ε, ε, προελήσεως ε, συνάδελφος σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Είμαστε όλοι τεχνοκράτες, εδώ ξέρουμε από αυτά. Εσείς είστε πολιτικοί, αλλά τα γνωρίζετε όλα αυτά τα στοιχεία. Σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία στην Τζέσικα και στον Τζέρεμι, ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρεται ε, σαν να ήταν ήδη κανονισμό το νέο αυτό εργαλείο. Θα ήθελα να το συνδέσω και να απαντήσω επομένως και στην κυρία Κέλμα με αυτόν τον τρόπο όσον αφορά το σύστημα ελέγχων. Εγώ αναφέρθηκα σε πέντε επίπεδα. Έχουμε ένα πρώτο επίπεδο, δεύτερο. Έχουμε το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πρέπει και αυτό να ελέγξει, το ε, Εθνικό Ελεκτικό Συνέδριο και το ε, ε, Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Έξι επίπεδα λοιπόν, έξι. Εγώ στην πρώτη μου παρέμβαση προσπάθησα με πολύ συνθετικό τρόπο να πω ότι η κατάσταση, η οικονομική και κοινωνική κατάσταση των ε, περιφερειών είναι τρομερή και είναι λες και έχει ξεσπάσει μια τρομερή πυρκαγιά και εμείς αντί να τη σβήσουμε προσπαθούμε να ελέγξουμε ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, εμείς προσπαθήσαμε λοιπόν να εγκαινιάσουμε διάλογο με την Επιτροπή χρησιμοποιώντας ε, τις ε, κοινέ checklists που έχουν εγκριθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μετά είχαμε και μία θετική εμπειρία των ε, κοινών ελέγχων Εθνικού ε, και Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ε, με τη σύμπτυξη αυτή φτάνουμε σε τρία επίπεδα ε, ελέγχου. Είναι και αυτά, και αυτά πολλά τα επίπεδα ελέγχου, αλλά παρόλα αυτά έχουν μειωθεί σε σχέση με τα πρώτα έξι. Ε, είναι μια εμπειρία που την έχουμε κάνει και έχει καλά αποτελέσματα και νομίζω ότι θα πρέπει να την αξιολογήσουμε στην παρούσα νομοθετική δέσμη, εν πάση περιπτώσει με κάποια σύσταση έστω εξ του Κοινοβουλίου, αν είναι δυνατόν, και αν είναι δυνατόν ακόμα και εξ των κρατών μελών. Äh, Ευχαριστώ για την προσοχή, για την παρατήρηση και τώρα ε, βλέπουμε ότι υπάρχει ο κύριος Τρίλιν και ο κύριος Μόλοφ που ζητούν το λόγο και, εσύ, και εσείς κύριε Λοχάιτ ε, έχετε ερωτήσεις. Ωραία. Ε, οι τρεις μυρογνώμονες για τον επόμενο γύρο ερωτήσεων. Πρώτα ο κύριος Τρίλινγκ. Ευχαριστώ πολύ. Το κατά πόσο θα πρέπει να εμφανίζεται ο κατάλογος των δικτών. Ναι, πιστεύουμε ότι οι στόχοι θα πρέπει να συνδυάζονται και να συνδέονται με τους θεματικούς στόχους. Και εδώ ε, στρέφομαι και θέλω να απαντήσω στον κύριο Μάρτιν αυτό που παρουσιάσαμε είναι το πιο ομαδοποιημένο επίπεδο. Ο ευρωπαϊκής στόχη λοιπόν που τίθενται σε, ευρωπαϊκό, ε, σε εθνικό επίπεδο επιθεματικών στόχων. Και εδώ βεβαίως σιγά σιγά ερχόμαστε και στο ερώτημα του κατά πόσον είναι ε, κατά πόσον οι δείκτες μπορούν να μας πληροφορήσουν ε, για την αποτελεσματικότητα των στόχων ή την αποτελεσματική εφαρμογή των στόχων. Και ένα βήμα παραπέρα ε, κράτη-μέλη τα οποία στα πλαίσια του πλαισίου απόδοσης μπορούν να θέσουν συγκεκριμένους στόχους ε, και κατά πόσον θα πρέπει να υπάρχουν ε, result indicators που θα συνδέονται με τους στόχους ε, αυτούς. The και βεβαίως θα πρέπει να βρούμε τον χώρο, το σημείο στο οποίο επιπλέον στόχοι, συγγνώμη, δείκτες αποτελέσματος μπορούν να καταδεικνύουν το επίπεδο της προτεραιότητας. Ε, στα πλαίσια του στόχου ε, θα έβλεπα εγώ και τα αποθεματικά και το θέμα των κυρώσεων επίσης, εάν και εφόσον δεν επιτευχθούν οι στόχοι από το ε, κράτος μέλλον. Επομένως, επιπλέον όθηση για επίτευξη των στόχων και κύρωση για περίπτωση μη επίτευξης. Και αυτό να εφαρμόζεται στις διάφορες περιοχές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος μόλο επόμενος. Ευχαριστώ. Αν κατάλαβα καλά, η ερώτηση αφορούσε το αν μπορεί το τοπικό επίπεδο να συνεργάζεται και να συνδυάζει τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής με ιδιωτική χρηματοδότηση. Και ποια είναι η δυνατότητα απορρόφησης των κονδυλίων. Σε ό,τι αφορά τις στρατηγικές, τις άτυπες, ε, την περιφέρεια αυτή, υπάρχει δυνατότητα διάφοροι δήμοι και κοινότητες να καταθέσουν ε, προγράμματα αξιόπιστα αποδοτικά με μεγάλη απόδοση και μπορούν να προσελκύσουν ιδιωτικά κεφάλαια από τις επιχειρήσεις. Και αυτό νομίζω μπορεί να έχει και καλύτερα αποτελέσματα και καλύτερη απορρόφηση των κονδυλίων. Αυτή τη στιγμή έχουμε προβλήματα με την ενιαία ε, αντιμετώπιση των ε, ε, προγραμμάτων και των έργων. Μπορεί να απορροφώνται τα κονδύλια, αλλά δεν υπάρχουν αποτελέσματα πάντα πρακτικά. Και αν ε, τα σχέδια ανταποκρίνονται και συνάδουν και με συμφέροντα ιδιωτικών επιχειρήσεων, μπορεί να είναι πιο ενδιαφέροντα τα αποτελέσματα. Έτσι μπορεί να γίνει καλύτερος σχεδιασμός πάντα με βάση την περιφερική τοπική ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λόχάιντε, πώς θα τα μεταφέρουμε αυτά στην πράξη με την απλοποίηση και τους ελέγχους. Ναι, και εγώ το ξέρω ότι δεν μπορούμε να πούμε στον κανονισμό, στο Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο να δεχθεί αυτά που έχουν ελέξει ή κάποια περιφερειακά ελεκτικά συνέδρια ή εθνικά. Και το αντίστροφο ισχύει. ποιος νομοθετεί σε εθνικό επίπεδο το κοινοβούλιο, αλλά υπάρχουν ε, διάφορα δικαιώματα διαφόρων επίπεδων. Δεν χρειάζεται να το πούμε σε αυτό τον κανονισμό, ε, αλλού όμως να λέμε ότι όταν έχει γίνει ο έλεγχος από τα περιφερειακά ελεγκτικά συνέδρια ή τα εθνικά, να μην χρειάζεται να ξαναγίνει και από το ευρωπαϊκό και μπορεί να προσκαλεί ε, τους ε, ενεχομένους εταίρους που έχουν υπογράψει αυτή τη σύμβαση εταιρικής σχέσης για να γίνεται με διαπραγμάτευση αυτή η διαδικασία και να το δέχονται. Δεν ξέρω στην πράξη πώς θα γίνει αυτό, αλλά θα έχει ένα αντίκτυπο. Σε, ε, ό,τι αφορά ένα άλλο θέμα για την καθάριση των λογαριασμών και ε, τις εκθέσεις που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μα γίνεται αυτό το πράγμα, να σας πω από την πράξη ενδεχομένω αν μου επιτρέπετε τι συμβαίνει και τι έχει σημασία. Πέρα από τα σχέδια και τα έργα που συνήθως είναι πολυετή και είναι σχετικό το αποτέλεσμα το τι μπορεί κανείς σε αιτήσια βάση να αναφέρει, αποκλίνουν τα χρονικά διαστήματα. Δεν είναι πάντα αιτήσεις οι εκθέσεις για το κλείσιμο των λογαριασμών. Θα ήταν καλό λοιπόν να έχουμε ενιαίες περιόδους αναφοράς για τους λογαριασμούς και είναι μεγαλύτερη διαφάνεια γιατί από χώρα σε χώρα διαφέρει αυτό, υπάρχουν αποκλήσεις και πάλι αυτό θα αύξανε και τη γραφειοκρατία και ενδεχομένως να ε, μην είχε και συγκρίσιμα αποτελέσματα. Ε, δεν ξέρω μήπως χρειάζεται ε, εκεί μια ενιαία προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις περιόδους αναφοράς. Ευχαριστώ. Ε, η κυρία Σρέτερ, βέβαια δεν εννοώ εσάς, έχουμε όμως 15 λεπτά. Ε, τρεις ερωτήσεις και μετά θα δώσουμε πάλι το λόγο στους ε, ειδικού. Σχετικά με το τελευταίο θέμα έχω μία πρόταση. Δηλαδή ε, όπου εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιπαρατίθεται εις την προσαρμογή των περιφερειακών ή εθνικών κανονισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαμε με αυτό να λύσουμε το πρόβλημα της αιρεσιμότητος. Αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο ελέγχθη σαφώς είναι ότι πρέπει να ρυθμίσουμε διαφορετικά τους δείκτες. Διότι έχουμε δείκτες οι οποίοι θεωρούνται κοινοί ε, και είναι δείκτες για τα μέτρα και όχι δείκτες για το αποτέλεσμα για τη μέτρηση του αποτελέσματος. Ρωτήσαμε γιατί υπάρχει αυτό, οπότε εγώ αναρωτιέμαι. Δεν είναι δυνατόν να εφαρμόσουμε την πρόταση του κυρίου Τρίλιχ, δηλαδή τουλάχιστον να υπάρχουν δείκτες που να είναι συνδεδεμένοι με το αποτέλεσμα, με τους στόχους. Οπότε ρωτάω πώς πρέπει να προχωρήσουμε. Πρέπει μόνο εκεί να υπάρχουν ευρωπαϊκοί δείκτες και στα άλλα επίπεδα όταν ε, να υπάρξουν απλώς ε, για ε, δείκτες για τις προτεραιότητες επενδύσεων ή αυτοί είναι δείκτες από τους οποίους μπορείτε να διαλέξετε, μπορείτε να προσανατολιστείτε. Μου φαίνεται πιο εφικτό και νομίζω ότι αυτό ακολουθεί και το πνεύμα του Γιάννη. Ε, σχετικά με το τι πρέπει να γίνει σε κοινοτικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο. Και ένα άλλο ερώτημα είναι το εξής. Αυτό το οποίο ε, αγνοήθηκε είναι ε, ο στρατηγικός έλεγχος περιβαλλοντολογικής αντοχής και αυτό πώς μπορούμε να το συνδυάσουμε με την επίδοση, την performance. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ο Μίχαλ Τόερεν είναι ο επόμενος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και για τους φιλελεύθερους θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές διότι τα σχόλια τα οποία κάνατε ε, είναι πολύ επιφυλακτικά σε σχέση με το στόχο τον οποίο έχουμε θέσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι ε, εδώ μιλάμε για την δημοσιονομική ρύθμιση την οποία διαπραγματευόμαστε με το Συμβούλιο και ρωτήθηκε εάν στα πλαίσια των ε, διαφόρων ταμείων το ποσοστό λάθος ε, ή αν είναι πολύ υψηλότερο. Κύριε Έλερ, δυστυχώς Όντως έτσι είναι. Μπορώ να σας το πω γιατί είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Το ποσοστό των σφαλμάτων είναι σημαντικότατο και γι' αυτό δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε έτσι. Γι' αυτό είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ας αλλάξουμε τους κανόνες και αν δεν θέλουμε, εάν θέλουμε να υπάρξει απλοποίηση που είναι κάτι που μας καίει εμάς σαν φιλελεύθερους, Οπότε πρέπει να δούμε αν μπορούμε να διευκολύνουμε τη ζωή μας, αλλά πρέπει να δούμε πώς θα επιτύχουμε τον ίδιο στόχο, το, τη μείωση ε, του ποσοστού των λαθών με τα νέα μέτρα. Οπότε σας ερωτώ, τι προτάσεις έχετε να διατυπώσετε συγκεκριμένα κατά τρόπον ώστε να έχουμε και ένα μοχλό διότι δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποχρεώσει τα εθνικά ηλεκτρικά συνέδρια ούτε τις εθνικές αρχές να τιμωρήσουν ούτε μπορούμε να θεωρήσουμε πρότυπο ε, τους δικούς μας κανόνες και αυτό ε, διακηρύσσεται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γι' αυτό πολύ σωστά είπε η κυρία Κρέλ υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις για το πόσο θα τα καταφέρουν τα κράτη-μέλη για να μην ζητούμε από, να, να, για να ζητούμε μεν από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να προβαίνει σε έναν έλεγχο για τον έλεγχο των ευρωπαϊκών πόρων αλλά σε, εθνικό επίπεδο να κάνει ο καθένας ε, τη δουλειά του στο χώρο του. Και αυτή είναι η ερώτησή μου, δηλαδή πώς θα το ρυθμίσετε εσείς και πώς θα το συζητήσετε με αυτούς που εφαρμόζουν τα μέσα και τα μέτρα στην περιφέρεια, στην περιοχή τη συγκεκριμένη. κύριος Γκάιερ. Υποστηρίζω τον πρόεδρο της Επιτροπής μου. Ναι, είναι πολύ υψηλότερο το ποσοστό σφαλμάτων. Παραμένει η αχίλιος πτέρνα του κοινοτικού προϋπολογισμού το Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εδώ είμαστε στο 7,7% πιθανό ποσοστό σφάλματος. Δηλαδή θεωρητικά μπορεί να είναι συν πλην 3% έτσι δεν είναι. Το ελεκτικό συνέδριο το παραδέχεται, αλλά 7,7% πιθανό περιθώριο σφάλματος είναι πολύ μεγάλο. Και κυρίε και κύριοι, το μεγαλύτερο ρίσκο και μεγαλύτερο κίνδυνο τη πολιτική συνογή αυτή τη στιγμή είναι να δανειστούν αυτό το ποσοστό σφάλματος ορισμένε κυβερνήσει και να πούν τα χρήματα δεν δαπανώνται με τρόπο σωστό και χρηστό, οπότε να μειωθούν τα ελεγκτικά συνέδρια συνεργάζονται στο βαθμό που αυτό γίνεται. Αλλά έχουν διαφορετικές πολλές φορές στρατηγικές και προδιαγραφές. Βλέπε τύπου <laughs> καθολικοί προτεστάντες και δεν μπορούν να συμφωνήσουν για το πώς θα φτάσουμε στην ε, ε, θέαωση. Ε, πάντως το συζητήσαμε αν μπορούν να συνεργαστούν. Έχω μια ερώτηση εγώ στους ειδικούς εμπειρογνώμονες. Έχετε ποτέ ψάξει για ποιο λόγο. Επειδή γίνονται πολλοί έλεγχοι. Παρόλα αυτά γιατί δεν πέφτει το ποσοστό σφάλματος. Γιατί ξέρουμε ακριβώς πού γίνονται τα λάθη. Και ο κύριος Γκαρτζούλο το είπε ε, για την περιφέρειά του και εντόνως ότι είναι έξι τα επίπεδα ελέγχου. και για να σας διορθώσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ελέγχει. Αντιπροσωπείες κάνουμε, εξεταστικές επιτροπές, ε, δηλαδή ελέγχουμε τα πράγματα επί τόπου, αλλά δεν ε, είμαστε ελεγκτικό όργανο. Αλλά η Ιταλία οφείλεται για το 20% των σφαλμάτων στην πολιτική συνοχή. Αφού είναι τόσο πολύ έλεγχη, γιατί παραμένει τόσο ψηλό το ποσοστό σφάλματος. Το έχετε κοιτάξει αυτό, το έχετε μελετήσει. Ε, ποια είναι τα προβλήματα τα διοικητικά που προκύπτουν. και οι ε, διατάξεις οι κοινοτικές με τις εθνικές δεν είναι συντονισμένες και φορτώνονται τα πάντα στην πλάτη του, τεχνικού, του τελικού δικαιούχου, ο οποίος δικαίως διαμετήρεται, αλλά δεν υπάρχει τελικά ε, αποτέλεσμα. Γκοτμάνης και Τσέλερ. Ευχαριστώ πολύ. Σε τελική ανάλυση, το θέμα είναι να δαπανώνει σωστά τα κονδύλια. Και ε, ζητώ από τους εμπειρογνώμονες και ε, θέλω να ρωτήσω τον Τζον Μπάχλερ, όπως ρώτησαν και τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμού. Κοιτώ τη διαφάνειά σας υπαριθμών 5. Λέτε ποιο είναι το πρόβλημα, αλλά δεν κάνετε προτάσεις. Και όπως λέμε, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Όλη αυτή η κατασκευή, πώς θα γίνεται η κατανομή, ο επιμερισμός των κονδυλίων, phasing out, phasing in, περιφέρειες, ε, υποκρισμένε. αυτό είναι στο παράρτημα 2 και μπορείτε να απαντήσετε. Τον κανονισμό 1083 ανοίξτε παράρτημα 2 και αυτά ορίζονται σαφώς. Ε, μπορεί να υπάρχουν ορισμένες πολιτικές προσαρμογές που έκανε τελευταία ώρα το Συμβούλιο για να ελέξει το σύνολο των πολιετών δημοσιονομικών προοπτικών. Σήμερα έχουμε μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακόμα και η Γενική Διεύθυνση ε, Περιφερειακή έχει περικόψει κονδύλια δισεκατομμύρια και στη σελίδα 62 του εγγράφου που σας δείχνω. Εσείς λοιπόν που είστε εμπειρογνώμων, έχετε καμιά ιδέα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρήσει τους σημερινούς μηχανισμούς που είχε υλοποιήσει και τους βάζει σε περιφέρειες υπομετάβαση τις καλώς ανεπτυγμένης και τις λιγότερο ανεπτυγμένης. Γιατί σήμερα είναι λευκή σελίδα το νομοθετικό πακέτο για τη συνοχή. Ο Δης γνωρίζει τι θα γίνει με τα 162 δισεκατομμύρια της λιγότερο ανεπτυγμένης περιφέρειας, πώς θα κατανεμηθούν, πώς θα επιμεριστούν εντός των περιοχών. 53,1 δις ας πούμε στις καλώς ανεπτυγμένες περιφέρειες. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο ερώτημα, ακριβώς το ίδιο. Εδώ μιλάτε για την οροφή, αυτό το κάπινγκ, κάπου να υπάρχει ένα το όριο. Και τι σημαίνει αυτό. Αντί για 4% ακούμε ότι θα είναι 2,5%. Αλλά στο παράρτημα 2 δεν λέει ούτε καν το 4% από 3,7 έπαιξε στο 3,2. Τι προτείνετε εσείς που τα ερευνάτε αυτά και τα ψάχνετε, ε, τι προτείνετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ρωτάμε την Επιτροπή και δεν έχει ιδέα σήμερα, ούτε καν προτίθεται να αλλάξει αυτούς τους μηχανισμούς. Τελικά όμως ο μεγάλος καυγάς μεταξύ των κρατών μελών δεν θα γίνει εδώ στην Επιτροπή μας, αλλά στο Συμβούλιο για το πώς θα κατανεμηθούν τα κονδύλια. Ευχαριστώ. Καλώς, ο συνάδελφος Τσέλερ και η κυρία Έρνς, πολύ σύντομα. Λοιπόν, εγώ δεν έχω τίποτα ενάντια στην αρμοδιότητα των ελεγκτικών συνεδρίων, αλλά ξέρω ότι τα ελεγκτικά συνέδρια έχουν και αυτά λόγο υπάρξεως ε, και κάνουν ελέγχους μέχρι να βρουν κάποιο λάθος, ακόμη και τυπικό. Οπότε αν δούμε το ποσοστό της διαπιστώσεως λαθών δεν μου λέει τι κρύβεται πίσω από το αποτέλεσμα διότι όταν πρόκειται για δημόσιους διαγωνισμούς, για δημόσιες προμήθειες είναι προφανώς προφανές ότι ε, όταν ε, πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μην υπάρξει κανένα λάθος και γι' αυτό χρειάζεται και ο έλεγχος από το ηλεκτρικό συνέδριο. Ευχαριστώ. Ε, η κυρία Ένστ, έχω δύο ερωτήσεις. Το ε, αφενός ε, μία συνάδελφος από την καμπάνια είπε ότι πρέπει να προσπαθήσουμε όταν μιλάμε για την ποικιλομορφία των περιφερειών να είμαστε πιο σαφείς και θα ήθελα να ξέρω για το απόθεμα αποδόσεως που είναι κάτι που δεν γνωρίζω δηλαδή ε, είναι ένα μέσο. Τι σημαίνει αυτό είναι κάτι το οποίο ενετάχθη την τελευταία στιγμή και ίσως μπορείτε εσείς κάπως να με διευκολύνετε να μου πείτε ε, τι εννοείτε όταν μιλάτε για επιδόσεις, για μέτρηση των επιδόσεων και ε, για απόδοση. Διότι είπατε εσείς ποσοστό λαθών 7,7%. Είναι ένας αριθμός και αυτός, εντάξει. Τι γίνεται όμως με τα πράγματα πραγματικά λάθη. Τι είναι τα λάθη. Ίσως η ε, ανεπαρκής απλοποίηση οδηγεί σε αύξηση των λαθών. Όταν μιλάμε για κάτι τέτοιο πρέπει να δούμε τι κρύβεται πίσω από τα σφάλματα. Και ε, γιατί χρειάζεται να υπάρχει πιστοποίηση. Δηλαδή ποιο γεγονός, ποια αιτία, ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χρειάζεται να υπάρχει υποχρεωτικά αυτή η πιστοποίηση, είναι θέμα ζωής και θανάτου. Δεν καταλαβαίνω, δεν έχω αυτή την εντύπωση. Λοιπόν, προτείνω τώρα επειδή ε, οι εμπειρογνώμονες δεν θα μπορέσουν να απαντήσουν σε όλα, εάν μείνει κάτι σε κρεμότητα να το λύσουν διμερώς. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιος θέλει να μιλήσει και να σχολιάσει για δύο λεπτά και τα υπόλοιπα μπορείτε να τα λύσετε διμερώς. Ο κύριος Βάχτλερ έχει ζητήσει το λόγο και θα ακολουθήσω τη σειρά έτσι μέχρι να τελειώσουμε. Ευχαριστώ. Δύο-τρία σημεία. Η ερώτηση της κυρίας Σουέτερ σχετικά με την στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση Στην έκθεσή μας ε, δεν υπάρχει δική αναφορά σε αυτό πάντως. Πιστεύω ότι στην πρόταση της Επιτροπής ε, υπάρχει ε, περιθώριο καλής εφαρμογής όσον αφορά τις προτάσεις για την αιρεσιμότητα. Ε, δηλαδή αυτή η αξιολόγηση μπορεί να είναι ένα μέσο βελτίωσης. Εάν βέβαια τα ετούμενα κριτήρια για την περιβαλλοντική αιρεσιμότητα καλύπτονται ε, στην πράξη, ε, και κατά πόσον θα χρησιμοποιηθούν ε, οι συζητήσεις και οι αξιολογήσεις ε, της αξιολόγησης μάλλον εξάντε και αν θα χρησιμοποιηθούν με αποτελεσματικό τρόπο αυτό έχει να κάνει με την στρατηγική ενσωμάτωση των οδηγιών κτλ. Νομίζω ότι ο κύριος Γκοντμάνης έκανε μια ερώτηση σχετικά με τους υπολογισμούς του προϋπολογισμού. έχουμε ξοδέψει πολύ χρόνο προσπαθώντας να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η κατανομή. Και βεβαίως κανείς μπορεί να κάνει κάποιες ε, εκτιμήσεις ε, σχετικά, αλλά παραμένουν σημαντικές άγνωστοι παράμετροι. Ας πούμε, μία βασική αρχή είναι ο, τρόπο με τον οποίο, ε, ο τρόπος με τον οποίο οι παρελθούσες χρηματοδοτήσεις ε, θα επηρεάσουν μελλοντικές χρηματοδοτήσεις. Επίσης, ε, η συνυπολόγηση των πραγματικών αναγκών των κρατών. Αυτές είναι, ε, αυτά είναι σημεία αρχής και ουσίας. Υπάρχουν κάποια προβλήματα σχετικά με τη διαφάνεια, δηλαδή ακόμα παραμένει ασαφές ποιες ποιες καταβολές θα γίνουν στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, επίσης ποια θα είναι η επιλογή σε μεθοδολογία ή ποιες θα είναι οι αρχές που θα διέπουν τη μεθοδολογία. Ε, θα ληφθεί υπόψη το, το παλαιό καθεστώς επιλεξιμότητας, ε, η τροποποίηση καθεστώτος ε, περιφερειών, το κατακεφαλήν, το ΑΕΠ, το κατακεφαλήν ΑΕΠ, εμείς έχουμε κάνει κάποιες συστάσεις και με βάση των οποίων χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια, κυρίως όσον αφορά τα κριτήρια των ε, πιο αναπτυγμένων και των ε, ε, μεταβατικών περιοχών. Όσον αφορά τώρα την οροφή, αυτό το κάπινγκ εισήχθη το θέμα του κάπινγκ εισήχθη αρχικά ως οροφία απορρόφησης και σας εξηγώ γιατί με βάση των προηγουμένων εμπειριών μας ξέραμε ότι υπάρχει ένα όριο ε, στο ποσοστό απορρόφησης, ε, το, ε, το, το maximum ποσοστό απορρόφησης που μπορούν να έχουν κάποιες περιοχές. Γι' αυτό είπαμε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτό το, το capping. Βεβαίως το σκεπτικό τώρα δεν είναι το ίδιο όσον αφορά την απορροφητικότητα γιατί μιλάμε πλέον για πολύ χαμηλότερα, πολύ μικρότερα ποσά. Ε, το πρόβλημα το οποίο μας απασχολεί εδώ, το αντίστροφο αποτέλεσμα δηλαδή που μπορεί να έχει, είναι ότι το κάπινγκ μπορεί να εφαρμοστεί σε σχέση με το ΑΕΠ, πράγμα που σημαίνει ότι χώρες οι οποίες ήδη δεν είναι πολύ εύρωστες ε, θα πάρουν ε, λιγότερη χρηματοδότηση, ενώ χώρες με πιο γερό ΑΕΠ θα δουν αύξηση και επομένως αύξηση και του, της οροφής αυτής του κάπινγκ. Ο επόμενος πολύ σύντομα, ο κύριος Τσούλεγ. Έγινε μια ερώτηση για την κρίση και πώς πρέπει να αλλάξει ο τρόπος χρηματοδότησης. Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος, ακόμα και στις σημερινές προτάσεις. Εκείνες οι περιφέρειες που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες ε, και δεν μπορούν ούτε να διαχειριστούν ούτε να απορροφήσουν ε, κονδύλια από διάφορες πηγές, θα αγωνιστούν και θα, θα ταλαιπωρηθούν για να τα εφαρμόσουν όλα αυτά και θα ξανάρθουμε μετά από πέντε χρόνια και θα διαπιστώνουμε στις περιφέρειες αυτές πάλι πολύ χαμηλή απορρόφηση. Και το θέμα είναι τι σκοπό έχει και τι σκοπό εξυπηρετεί η περιφερειακή πολιτική τελικά και η πολιτική συνοχής. Για τους δείκτες, κάτι που μου λείπει από τη συζήτηση είναι η σύνδεση των στόχων της επίδοσης και των δικτών αποτελέσματος. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας μια ξεκάθαρη ιδέα για το ποιο είναι το μοντέλο πολιτικής που κρύβεται από πίσω. Ας πούμε, οι δαπάνες και τα κονδύλια σε μια συγκεκριμένη πολιτική Πού οδηγούν, τι θέλουμε να έχουν ως αποτέλεσμα. Και αν δεν διευκρινίσουμε αυτή τη διαδικασία, από μόνοι τους οι δείκτες αποτελέσματος θερούνται εννοήματος. Γιατί δεν μπορούμε να τρίσουμε κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το συνδέσουμε ξανά με τη δαπάνη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τρίλινγκ. Ευχαριστώ πολύ. Διάφορα επίπεδα δικτών. Μάλιστα. Νομίζω ότι σε επίπεδο θεματικών στόχων και σκοπών πραγματικά χρειαζόμαστε δείκτες που να δείχνουν τις επιδόσεις και των κρατών μελών και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν πληρώσει τους στόχους τους στα κράτη. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και για να υπάρξει ε, λεπτή ε, σύγκριση χρειάζονται πιο ειδικοί δείκτες που και μάλιστα μέχρι το περιφερειακό επίπεδο, να μην σταματούν στο εθνικό. Η στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση τώρα είναι το μόνο νομικά κατοχυρωμένο εργαλείο που θα εξασφαλίσει τη συνοχή των προγραμμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται σε αυτό σε σύνδεση με άλλες δοκιμές για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα Εκ των προτέρων όμως είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο να γίνεται από πριν. Γι' αυτό και η εκ των προτέρων αιρεσιμότητα για να βεβαιωθούμε ότι συμμορφούνται προς το SEA. Αλλιώς είναι πολύ αργά. Τώρα αρχίζει η προγραμματική περίοδος και έχουμε πήραμε χώρες που χωλένουν ε, στην εμπειρία τους ε, και στην τελευταία προγραμματική περίοδο δεν είχαν επιτύχει πάρα πολύ και τελικά αυτό το στοιχείο αποδείχθηκε άχρηστο το, η στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση λοιπόν. Θα πρέπει να εφαρμοστεί ήδη από τώρα η οδηγία αυτή και να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση. Και ένα άλλο στοιχείο που θα ήθελα να αναφέρω εδώ είναι το πώς ενέχονται οι διάφοροι εταίροι στο προγραμματισμό, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση και τον έλεγχο για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η απόδοση όλων των ενδιαφερομένων θα πρέπει ο κώδικας συντολογίας που προβλέπεται να ε, δείχνει σαφώς τα ωφέλη Ποιες είναι ελάχιστες προδιαγραφές και βέλτιστες πρακτικές που θα μπορούσαν να ε, υιοθετήσουν σε εθνικό επίπεδο τα κράτη. Ευχαριστώ πολύ. Τέλειωσε ο χρόνος μας. Δυστυχώς έχουμε χρόνο μόνο για έναν εμπειρογνώμονα. Συνεννοηθείτε μεταξύ σας ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μιλήσει. Σχετικά με το θέμα των δικτών, απλούστατα θα ήθελα να πω ότι υπάρχει δυνατότητα να το επεξεργαστούμε και να σας πούμε τι δεν έχουμε κάνει και τι συνέβη όπου το εφαρμόσαμε. Ε, σχετικά με το ποσοστό λαθών και των σχετικών στοιχείων αναρωτιέμαι εάν η δημιουργία ενός, μιας νέας αρχής ε, θα μειώσει το ποσοστό σφαλμάτων ή θα κοστίσει υπερβολικά σε σχέση με το αποτέλεσμα. Οπότε ε, δεν θα πρέπει να μιλάμε για το κόστος σε σχέση με τα λάθη αλλά να υπάρχει εποπτεία στα διάφορα επίπεδα. Και τέλος ίσως θα ήταν πολύ πιο απλό αν μπορούσαμε να ε, κάνουμε τους ελέγχους από κοινού. Οπότε θα ε, λυνόντουσαν πολλά τα προβλήματα διότι θα βλέπατε ότι αν γίνει ένας ε, έλεγχος σε μία αρχή δεν παίζει κανένα ρόλο αν δώσουμε δύο περισσότερα εθνικά στοιχεία ή όχι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για όλους αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν στη συζήτηση αυτή και σας ευχαριστώ και εν ονόματι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι σήμερα μάθαμε πολλά πράγματα σχετικά με τη διεκπαιρέωση ή την προβλεπόμενη διεκπαιρέωση ε, του προγράμματος ε, ε, συνοχής και τώρα ερχόμαστε σε μία έκθεση που θα παρουσιάσει ο εισηγητής Γιώχιμ Τσέλερ αλλά με τη σύμπραξη με τον κύριο Μισελ Ντελμπάρ εισηγητή της Επιτροπής των περιφερειών και θα μιλήσουν για την τροποποίηση του κανονισμού ο αριθμός 1082 ε, του 2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας όσον αφορά την αποσαφήνιση, απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και εφαμοργής αυτών των ομίλων. Είναι ένας μακρύς τίτλος αλλά φαντάζομαι ότι γι' αυτό και τα λόγια του κυρίου Ντελμπάρ τώρα, ο οποίος θα παρουσιάσει το θέμα εν ονόματι της Επιτροπής Περιφερειών, θα είναι πολύ σημαντικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη ε, και από τα μέλη του Κοινοβουλίου γιατί εγώ δεν είμαι ο συγγραφεύς αυτής ε, της ποιητικής ε, συλλογής που και τελεί τίτλο, καθήκον ε, τίτλου εδώ πέρα. Λοιπόν, η πρόταση τροποποίησης ε, που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οδήγησε στην ε, έκθεση αυτή ε, που θέλει να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας, ΕΟΕΣ. Δεν είναι ένα απολύτως νέο εργαλείο. Ε, υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά πρέπει να επιστήσω την προσοχή των μελών του Κοινοβουλίου επί του σημείου ότι υπάρχουν 23 ΕΟΕΣ που έχουν ήδη συσταθεί που, όπου συμμετέχουν πάνω από 550 οτά σε 15 διαφορετικά ε, ε, κράτη και που ε, αφορούν πάνω από 22 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Υπάρχουν επίσης κι άλλες οι οποίες βρίσκονται καθοδόν προς την υλοποίησή τους. Επομένως δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι μια πραγματικότητα η οποία υφίσταται ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να υπενθυμίσω ότι η αναθεώρηση, η τροποποίηση μάλλον του κανονισμού δεν συνδέεται με τα διαρθρωτικά ταμεία. Παρουσιάζονται ε, στο, στην ίδια ομάδα στοιχείων, αλλά πρόκειται εδώ για ομίλους που δεν χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και ούτε από τα διορθωτικά ταμεία. Γι' αυτό λοιπόν η Επιτροπή Περιφερειών υπογραμμίζει την σημασία αυτού του κανονισμού που δεν έχει επίπτωση στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και ζητά άμεση έγκριση του συνόλου της δομοθετικής δέσμης των μέτρων για την πολιτική ε, για την συνοχή στην οποία συμμετέχει ο κανονισμός αυτός. Δυστυχώς όμως πρέπει να πω η παρούσα προεδρεύουσα του Συμβουλίου φαίνεται ότι δεν βρίσκεται στο ίδιο μήκος ε, κύματος. Δεν θέλει να βγάλει, να αποσυνδέσει ε, αυτό τον κανονισμό για τις ΕΟΕΣ ε, από το υπόλοιπο νομοθετικό πακέτο και φοβούμε ότι θα αναβληθεί διαρκώς ε, και βλέπε να αναβληθεί έως τις ελληνικές καλένδες ή μάλλον τις κυπριακές καλένδες, μια και αυτή είναι η επόμενη προεδρία. Εν πάση περιπτώσει ευελπιστώ κύριε Πρόεδρε ότι οι ευρωβολευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενδεχομένως θα μας βοηθήσουν έτσι ώστε να γίνει δεκτός ο κανονισμός αυτός. Ε, μία νέα ε, μορφή του κανονισμού βάσει της τροποποίησης αυτής ε, θα μπορούσε να δώσει νέα όθηση στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας και να ενδυναμώσει επομένως την συνεργασία μεταξύ των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την άποψη της Επιτροπής των Περιφερειών η τροποποίηση δεν ε, ε, δημιουργεί κανένα πρόβλημα στον, ε, στον υφιστάμενο κανονισμό. Απλώς ενδυναμώνει βάση του κανονισμού την, τον όμιλο εδαφικής συνεργασίας και επιβεβαιώνει και τον ρόλο της Επιτροπής των Περιφερειών στη δημιουργία και την προώθηση των ε, ΕΟΕΣ. Υπενθυμίζω τελειώνοντας ότι η Επιτροπή Περιφερειών προτείνει ε, να υπάρχει μια περιοριστική συλλητατική ερμηνεία των δυνατοτήτων απόρριψης ε, του αιτήματο για δημιουργία Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας. Επίσης ε, να ζητούμε να μην εμφανίζεται στον κανονισμό ε, ε, να μην υπάρχει η ανάγκη σε συγκεκριμένων νομοθετικών ε, προτάσεων. Εννοώ δηλαδή ότι να υπάρχει διοικητική απλούστευση και επίσης και οι όμιλοι ή οι οργανισμοί οι οποίοι ασχολούνται και συμμετέχουν στον όμιλο εδαφικής συνεργασία να θεωρούνται ε, κοινή ωφελίας. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό κυρίως σε ε, διασυνοριακές συνεργασίες. Ε, επίσης ε, στην επίσημη εφημερίδα ε, θα ε, πρέπει η ίδια η Επιτροπή Περιφερειών να δημοσιεύει την την ε, δημιουργία του ομίλου εδαφικής ε, συνεργασίας, τον οποίο θα οφείλει η ίδια η Επιτροπή Περιφερειών να παρακολουθεί. Νομίζω ότι χρειάζεται εδώ, αγαπητέ Πρόεδρε, να συγκλίνουν οι απόψεις μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να έχουμε μια ε, τεχνική βοήθεια, μια ταύτιση απόψεων για ένα θέμα το οποίο μπορεί να είναι σημαντικό για την εδαφική συνεργασία, χωρίς να έχει όμως καμία επίπτωση στον προπολογισμό. Πιστεύουμε ότι με, μέσω της τροποποίησης του υφισταμένου κανονισμού 1082 του 2006 μπορούμε να μεταδώσουμε τον ιό του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας ε, και στα άλλα θεσμικά όργανα ε, και επομένως ε, να βοηθήσουμε τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας να απλωθούν και πέραν των εθνικών συνόρων. Προ Επίσης ε, εμείς ε, ζητούμε ε, να υπάρχει η πρόσβαση του ομίλου συνεργασία συνεργασίας και σε άλλες, να διευρυνθεί μάλλον η δράση των ομίλων αυτών και πέραν των ορίων της πολιτικής σύνοχης. Αυτά ήθελα να σας πω και ευελπιστώ ότι η φιλοσοφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμεριστεί την φιλοσοφία της Επιτροπής Περιφερειών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Τσέλε, και μετά στους συντονιστές, στο βαθμό που θα είναι παρόντες, για να ακούσουμε τις απόψεις Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Ντελμπάρ, καθώς επίσης και την Επιτροπή Περιφερειών, που με τόσο σθένος ε, είναι προσιλωμένη στην υπόθεση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας αυτό είναι ένα μέσο που έχει προέρθει από τις ίδιες περιφέρειες, είναι τέκνο των περιφερειών. Και το σημειώνω ότι ο ιός αυτός είπατε θα πρέπει να είναι μεταδοτικός. Ήδη έχει κολλήσει κι αλλού. Είναι σχετικά νέο ε, νομικό μέσο. Υπάρχουν ήδη πάνω από 20 τέτοιοι όμιλοι εδαφικής συνεργασίας και πολλές περιφέρειες είναι σε λίστα αναμονής και θέλουν να συστήσουν ένα τέτοιο όμιλο εδαφικής συνεργασίας. Και νομίζω ότι είναι και απαραίτητο αυτό το μέσο για να ε, μεγαλώσει και να συνεργαστεί η Ευρώπη και να έχουμε μια κοινή πορεία. Γιατί στα κράτη-μέλη, παραμεθόριες περιοχές, οι ε, ακραίες περιοχές είναι εκείνες που κοινωνικά και οικονομικά υστερούν. Δεν είναι τόσο καλά ανεπτυγμένες ακόμα όσο τα κέντρα στην Ευρώπη. Και η Ευρώπη για να προχωρεί και να αναπτύσσεται μαζί θα πρέπει να ξεπεράσει τα σύνορα και ιδιαίτερα τα σύνορα των κρατών μελών. Πολλές από τις παραμεθόριες περιοχές το έχουν αναγνωρίσει και θέλουν να το εξασφαλίσουν και νομικά. Εξού και η όμιλη εδαφική συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω ανταποκρίθηκε πολύ σωστά σε αυτό, ε, διότι διεύρυνε τον ισχύοντα μέχρι σήμερα κανονισμό και δεν ε, περιορίζει τη ρισκή του μόνο εντός των σύνορων τη Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με τα εξωτερικά σύνορα, με περιφέρειες, το έχει επεκτείνει σε γειτονικά κράτη-μέλη για να μπορέσει να ελοποιηθεί περιφερειακά και να υποστηριχθεί η πολιτική γειτονία. Και το φάσμα των θεμάτων επίσης για του ομίλους εδαφικής συνεργασία, έχει διευρυνθεί δημόσιες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ιδρύουν τέτοιους ομίλους ή να συμμετέχουν σε τέτοιους ομίλους εδαφικής συνεργασίας και διάφορες πολιτικές ενίσχυσης θα πρέπει να ε, μπορούν να συνδυάζονται σε έναν ενιαίο όμιλο. Οι δυσκολίες τώρα ποιε είναι. Είχε την καλοσύνη να τις επισημάνει και αυτές ο κύριος Ντελμπάρ. Νομίζω ότι στις ίδιες περιφέρειες αλλά και στην Επιτροπή Περιφερειών θα είναι λιγότερες μάλλον δυσκολίε. επιφυλάξει, διατηρούν τα κράτη-μέλη και επίση δεν είναι και πάρα πολύ γνωστό αυτό το μέσο. Ούτε καν συνάδελφοι στο κοινοβούλιο δεν το γνωρίζουν ε, επαρκώς. Για να μην μιλήσω για άλλε ε, ε, θέσεις πέραν της Επιτροπής Περιφερειών. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει γνωστή αυτή η προσπάθεια και να προωθείται η εργασία τους στη διασυνοριακή συνεργασία. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό το μέσο κατά την άποψή μου. Για τις πέντε άλλες προτάσεις σε σχέδια κανονισμού πρέπει να πω ότι εδώ έχουμε συνέχιση και διεύρυνση, δεν είναι αναδιατύπωση του κανονισμού. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε εδώ ότι αυτό που κυριαρχεί εδώ δεν είναι τα χρήματα, δηλαδή η χρηματοδότηση των ταμείων συνοχής και των διαστατικών ταμείων, αλλά η επιτάχυνση της εργασίας. Επειδή δεν έχει να κάνει με χρήματα, λοιπόν, αυτός ο κανονισμός θα μπορούσε να προχωρήσει πιο γρήγορα. Λυπάμαι που η παρούσα Προεδρία του Συμβουλίου δεν έδραξε αυτή την ευκαιρία. θα πρέπει να αγωνιστούμε και εμείς για να πείσουμε πολλούς σε πολλά μέτωπα ακόμα. Σημειώνω τις παρατηρήσεις σας και τις προτάσεις σας για βελτίωση ε, του παρόντος κανονισμού για τον όμιλο εδαφικής συνεργασίας. Είναι σκόπιμα αυτά που λέτε και από εδώ και πέρα αρχίζει η πραγματική δουλειά, όχι τόσο πολύ εδώ στη δική μας Επιτροπή, γιατί οι συνάδελφοι εδώ είναι πεπισμένοι για την αναγκαιότητα και για τη χρησιμότητα αυτού του μέσου εκεί που θα χρειαστεί εφαρμογή και στους άλλους ε, κανονισμούς και στα άλλα σχέδια κανονισμών και στις υπόλοιπες στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και απέναντι στα κράτη-μέλη βεβαίως, όπου θα χρειαστεί να κάνουμε δουλειά. Ε, ε, προσβλέπω στη δική σας υποστήριξη και την Επιτροπή της Περιφερειακής Επιτρο... Συγγνώμη, τη στήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής την έχετε και εσείς σίγουρα και είναι δεδομένη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σμόλκοβα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά την περασμένη φορά. Ε, θα ήθελα και πάλι να επενέσω ε, τον κύριο Ντελμπάρ και να αποτίσω φόρο τιμή στο έργο της Επιτροπής Περιφερειών. Συμφωνεί το Κοινοβούλιο με αυτά που λέτε. Και πάλι δεν καταλαβαίνω γιατί έχει προβλήματα η ιδανική προεδρία. Κανονικά, αν εφαρμοστεί εγκαίρως αυτός ο κανονισμός θα έχει και πολλά πλεονεκτήματα για τη συνεργασία μας. Το ξέρω ότι υπάρχει έλλειμμα πληροφόρηση και στα κράτη-μέλη και μια ανησυχία ότι δεν θα συμμετάσχουν αρκετοί σε αυτή τη μορφή εδαφική συνεργασία στον όμιλο εδαφική συνεργασία. Όποιο το ακούει για πρώτη φορά τρομάζει, γιατί φοβάται ότι είναι πολύ μεγάλη διοικητική επιβάρυνση και γραφειοκρατία. Ωστόσο, ο κανονισμό αν το διαβάσει κανεί, δείχνει ότι χρειάζεται θάρρο και μπορούμε να προχωρήσουμε προ την κατεύθυνση αυτή χωρί να έχουμε επιφυλάξεις. Και για τι δημόσιε επιχειρήσει θα ήταν πολύ μεγάλη η ωφέλεια και το πλεονέκτημα. Το Κοινοβούλιο, είμαι σίγουρη, δεν έχει κανένα πρόβλημα, το έχουμε συζητήσει ήδη αυτό το θέμα, αλλά όπως είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως, θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και να τη συσφίξουμε. Τελευταίος ο Φρανσουά Αλφονσί. Ευχαριστώ. Για να ακολουθήσω την κατεύθυνση των προλαλισάντων, Όντως αυτό αποτελεί μια μεγάλη ε, ε, πρόοδο και πολύ καλή ε, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ένας τρόπος να δώσουμε με μια νέα όθηση στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Υπάρχει τεράστια ανταγωνιστικότητα η οποία ε, αναπτύσσεται ε, και βλέπουμε ότι ε, ακόμη και περιοχές που ήταν γεωγραφικά πολύ κοντινές είχαν μεγάλα, μεγάλες διαφορές στην ανάπτυξή τους. Τώρα βλέπουμε λοιπόν ότι εάν δεν, ακόμη και αν δεν πρόκειται για έναν κανονισμό φεντέρ ή εδαφικό εδαφικής ε, συνεργασίας αυτό που μας προτείνουν είναι τόσο λογικό ώστε δεν θα πρέπει να ε, δημιουργήσει προβλήματα και ε, θα μπορούσαμε να δώσουμε μία νέα όθηση σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ζητώ παρακαλώ τον κύριο Ντελμπάρ να κάνει μερικά σχόλια. Μάλλον με συγχωρείτε, είσαστε κι εσείς, δεν σας είχα δει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Θέλω να ε, συγχαρώ τον κύριο Τσέλερ αλλά και τον κύριο Ντελαμπάρ για το ε, εξαιρετικό ε, υλικό το οποίο πόνισε διότι Εν συντομία αυτή, αυτός ο όμιλος δίνει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες και οι τοπικές αρχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη νέα δυνατότητα και όταν θα έχει ολοκληρωθεί και ψηφιστεί ο κανονισμός αυτός η κατάσταση θα απλοποιηθεί διότι υπάρχουν 79 διαφορετικοί οργανισμοί για να που εμπλέκονται εις ε, την ε, ψήφιση ε, του κανονισμού αυτού στα 27 κράτη-μέλη. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα one-stop shop. Αλλά τι μας απασχολεί και αυτό ελέγχθη και μάλιστα σαφέστατα το θέμα της απλοποίησης. Εκεί κάτι πρέπει να κάνουμε. Και τέλος βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη ζητούνται να εφαρμόσουν τα μέτρα και να τα εναρμονίσουν διότι δεν είναι δυνατόν πλέον να υπάρχει μία αυθαίρετη ερμηνεία και η διοίκηση θα πρέπει να αντιληφθεί ότι μη ένα τέλος δεν έχει σχέση με την ε, περιφερειακή ε, πολιτική δεν πρόκειται για ένα τέρας το οποίο ε, θα δημιουργηθεί και θα χρειαστεί τεράστια μέση αν αυτό γίνει αντιληπτό και υλοποιηθεί τότε θα μπορούν να λαμβάνουν οι φάση σε τοπικό επίπεδο και ελπίζουμε ότι το μέσο αυτό θα μπορέσει να μας είναι πολύ χρήσιμο. Η Μαρή Τερέζ Σάντσες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοί μου. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Ιωάχιμ Τσέλερ για ε, την ακρίβεια των παρεμβάσεών του και να τονίσω πόσο συμφωνώ ιδιαίτερα με αυτή την ε, ιδέα της μονοαπευθυντικής σειρίδας το One Stop Shop που πρότεινε. Υπάρχουν ακόμα περιθώρια για πρόοδο στη διακυβέρνηση και στη διαχείριση ε, ανάλογα με το διαφορετικό επίπεδο αρμοδιότητας, ανάλογα με τη χώρα, καμιά φορά πραγματικά είναι γελίες οι καταστάσεις, ευτράπελες που ζούμε, ε, ιδιαίτερα ε, ως προς το προσωπικό που έχουν διαφορετικό καθεστώς οι εργαζόμενοι. Για το άλλο λοιπόν αυτό της διακυβέρνηση τοπική φορείς, στη δράση τους ή στην επικράτειά τους δεν μπορούν να αποκλείονται από τη διαχείριση ενός ομίλου εδαφικής συνεργασίας και δεν θα με διαψεύσετε εσείς κύριε Ντελπάρ. Εγώ το ζω επί τόπου. Είναι τεράστιο το πρόβλημα και κινδυνεύουν να χαθούν και κάποιες δομές που ήδη έχουν οικοδομηθεί εκεί ε, στον Όμιλο Εδαφικής συνεργασία. Δεν θα πρέπει να χάνουμε την επαφή μας με την πραγματικότητα στη διαχείριση και διακυβέρνηση αυτών των δομών. Ευχαριστώ. Μισελ Ντελμπάρ, έχετε το λόγο για να ολοκληρώσετε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, δεν θα επανέλθω εν λεπτομερία γιατί οι παρεμβάσεις όλων των μελών της Επιτροπής, που που πήραν τον λόγο ε, συγκλίνουν στην ανάγκη επιτάχυνσης γρήγορων διαδικασιών όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφική Συνεργασίας και επομένω ε, πρέπει να στραφούμε όλοι μαζί προ το Συμβούλιο για να πούμε ότι δεν χρειάζεται να συνδέσετε τον κανονισμό για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφική με την νομοθετική δεσμή στο πλαίσιο τη πολιτική για τη συνοχή ε, διότι δεν υπάρχει τέτοιος λόγος. Ε, τέλη Μαρτίου έχουμε διαθεσμική διοργανική συνεργασία όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας και ε, ευελπιστώ ότι ε, μπορούμε με αυτή την ευκαιρία να εκφράσουμε αυτές τις συγκεκριμένες απόψεις όσον αφορά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Περιφερειών. Να πω δε στην κυρία Σάντσε Σμιτ ότι η ΕΟΕΣ ήταν η καλύτερη δομή ε, για την θέση σε εφαρμογή ε, των ε, δομών πολλαπλής διακυβέρνησης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γιωακήμ, θες να ξαναπάρεις το λόγο. Όχι. Επομένως μπορούμε να ολοκληρώσουμε το σημείο αυτό και να πάμε στο σημείο 14 ε, της ε, ημερησίας διατάξεως. Είναι η έκθεση της Ρίκα Μάνερ, Συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στην επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Εντατικής Συνεργασίας. Δεν έχουμε εδώ εκπροσώπηση από την Επιτροπή των Περιφερειών. Θα σας δώσω επομένω άμεσα το λόγο έτσι ώστε να παρουσιάσετε το θέμα σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι κρίμα ειλικρινά που δεν παρευρίσκεται ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Περιφερειών για να το συζητήσουμε μαζί του. Γιατί ακριβώς ε, αν έχουμε υπόψη μας το χρονοδιάγραμμα τώρα είναι η στιγμή να συζητήσουμε μαζί τους. Δεν ξέρω μήπως ήταν εδώ το πρωί, εν πάση περιπτώσει. Κρίμα. Ελπίζω αυτό να μην σημαίνει ότι δεν θα συνεργαστούμε με την Επιτροπή Περιφερειών. Εμένα με ενδιαφέρει πολύ η θέση τους, όλους φαντάζομαι. Εχθές σας έστειλα ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, email, με το κείμενό μου. Το έγγραφο εργασίας, δεν θα σας το διαβάσω σε λεπτομέρειες, το έχετε στα χέρια σας. Απλώς θέλω να αναφέρω μερικά σημεία που αν θέλετε θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Αναφέρω το θέμα του προπολογισμού πρώτα απ' όλα. Ήδη το συζητήσαμε λίγο. Αυτό έχει να κάνει με το άρθρο 84 θα το συζητήσω και με τον εισηγητή για τον κανονισμό. Είναι σαφές ότι αυτό το θέμα το 3,4% αντί για 8% που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θέμα που πρέπει να συζητήσουμε για να δούμε αν μπορούμε να ε, έχουμε και γνώμη ως κοινοβούλιο και να μπει σε αυτή την έκθεση. Γνωρίζουμε ότι η συζήτηση για τον προϋπολογισμό πάντα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και τελικά, αν ζητήσουμε 7% μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα επιρροής και να ευδοκιμήσει η πρότασή μας. Είναι καλύτερο αυτό από εκείνο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη συνέχεια, Έχουμε και το μέσο ευελιξίες. Από προηγούμενα έτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα δεν το επανυποβάλλει, δεν το προτείνει. Γιατί λέει ότι δεν έχει απορροφηθεί το μέσο ευελιξίες στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο και εντάξει. Γιατί αυτό που το βρήκανε. Τα μισά κράτη-μέλη το έχουν χρησιμοποιήσει. Άρα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην πρόταση. Εμείς θεωρούμε ότι θα υπάρξει αύξηση της απορρόφησης και της ε, χρήσης του μέσου ευελιξίας και θα πρέπει οπωσδήποτε να μπει στην πρόταση. Προτείνω λοιπόν να επαναφερθεί, να επανέλθει, 15% ε, είναι ε, το έχω συζητήσει και με τους κοιόδης ηγητές και το θέμα της συγχρηματοδότησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 75% για όλες τις χώρες. Συμφωνώ. Δεν ξέρω αν θέλετε να συζητήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες προσαρμογής του ποσοστού. Σε γενικές γραμμές συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να το συζητήσουμε με τον εισηγητή της Επιτροπής Περιφερειών και τον, και τον ε, εισηγητή για τον Γενικό Κανονισμό, ο οποίος αυτή τη στιγμή απουσιάζει, αλλά θα το δούμε. Και έχω μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το άρθρο 11 του κανονισμού. Εκεί ε, δεν γίνεται λόγος για το ETC. E Αυτό τι είναι τώρα, το έχετε σκεφτεί ή όχι. Οι θεματικές στοχεύσεις. ETC είναι η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία. Είναι πολύ δύσκολο, το γνωρίζω, αλλά γιατί δεν το έχετε εντάξει εκεί. Και θα ήθελα να προτείνω στους κοιόδης ηγητές, αν μπορούμε, να συμπεριλάβουμε τρία υποχρεωτικά θέματα στην ε, συνεργασία και ένα προαιρετικό. Να επιλέγει το κράτος μέλος το τέταρτο θέμα. Δεν ξέρω τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό. Το έχετε εξετάσει, υπάρχει κανένα συγκεκριμένο πρόβλημα που θα απέκλειε κάτι τέτοιο. Τρία υποχρεωτικά, ένα προαιρετικό. Για τις μακροπεριφέρειες τώρα. Το κράτος μέλος είναι εκείνο που επιλέγει τα τέσσερα θέματα, λέτε. Εγώ διερωτώ με τι γίνεται με τις μακροπεριφέρειες. Θα πρέπει να περιοριστούμε σε αυτά τα τέσσερα θέματα. Αν γίνει αυτό, και πάλι περιορίζουμε αρκετά τις στρατηγικές της μακροπεριφέρειας. Γι' αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε και να το διευκρινίσουμε. Συνεχίζω. Το θέμα της απλοποίησης. Στον κανονισμό περιλαμβάνεται η δυνατότητα να, ε, συνένωσης των αρχών εποπτείας και ελέγχου. Εντάξει, καλό βήμα μου φαίνεται αυτό και για την εδαφική συνεργασία. Στη συνέχεια το flat rate, ο ενιαίος συντελεστής. Συμφωνώ. Ακριβώς, είναι χρήσιμο για την εδαφική συνεργασία. Είναι 50% αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε και αυτό το ποσοστό, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν μικρά προγράμματα που περίπου το μισό του κόστους είναι το διοικητικό κόστος. Ε, σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να μιλήσουμε για αύξηση του 50% που βλέπετε ως ενίο συντελεστή σε αυτό το flat rate. Και τέλος, για τη συγχρηματοδότηση σε όλους τους κανονισμούς, το είπα και για το γενικό κανονισμό και το έθεσε υπόψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί στο άρθρο 88 δεν αναφέρεστε στην εδαφική συνεργασία. Ω στόχο ακριβώ συνεργασία μεταξύ των διαφόρων κανονισμών. Γιατί έχει φύγει αυτό, γιατί το έχετε παραλείψει. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία εκεί να ενταχθεί, γιατί ακριβώ. η συνεργασία των διαφόρων τοπικών φορέων, εδαφική συνεργασία είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχει πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Πάρα πολύ... Γρήγορα λοιπόν αυτά ήταν τα βασικότερα σημεία που ήθελα να θέσω υπόψη. Βεβαίω υπάρχουν και λεπτομέρειες και πολύ πιο τεχνικά ζητήματα. Σας προτείνω όμως να αφήσουμε τα τεχνικά ζητήματα στην άκρη για αργότερα. Προς το παρόν να μην ασχοληθούμε με αυτά. Γνωρίζω ότι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου θα ψηφιστεί τον οι τροπολογίες εδώ στην Επιτροπή μας και μετά δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να πάμε στην Ολομέλεια το δεύτερο ήμις του Μαΐου. Εν πάση περιπτώσει είμαι στη διάθεσή σας ε, για τα σχόλιά σας, προτάσεις, ό,τι άλλο θέλετε. Ευχαριστώ. Φαντάζομαι ότι οι σκιώδες θέλουν να μιλήσουν. Μαρή Τερές. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια γιατί η έκθεσή της πραγματικά βρήθη καλών ε, στοιχείων, εργάστηκε με μεγάλη ακρίβεια ε, και δεν πρέπει να λησμονούμε όταν συζητούμε το μέλλον της πολιτικής συνοχής ότι η εδαφική, ευρωπαϊκή διαφυγική συνεργασία μπορεί να είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο απέναντι στην ε, κρίση. Είμαι πεπισμένη και το έχω επανειλημμένα πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λειτουργήσει μονάχα εάν ενισχύσει αυτά τα σημεία ένωσης ε, και εάν ε, μπορέσει να ενισχύσει τη διασυνοριακή ε, συνεργασία. Θα θίξω κάποια στοιχεία τα οποία θίξει ήδη και η κυρία Καμάνερ. Προϋπολογισμός. Τι προϋπολογισμό, ποιο προϋπολογισμό θέλουμε. Ε, και ζητούσαμε και στην έκθεση 7% ε, για την πολιτική συνοχής. Ε, η Κομισιόν ζητάει 3,48 ε, και νομίζω ότι αν είμαστε συνεκτικοί πρέπει να διατηρήσουμε το επίπεδο που είχαμε ζητήσει πριν. Ε, Παρ' όλα αυτά παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα. Θα επιτύχουμε την επιπλέον χρηματοδότηση στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής. Εάν ζητήσουμε απλά αύξηση θα πρέπει να ζητήσουμε προηγουμένως τη γνώμη των συναδέλφων της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Θα πρέπει πάντως να είμαστε φιλόδοξοι. Μία ερώτηση Προ προς την Επιτροπή θα ήθελα τώρα ε, όσον αφορά την ε, κατανομή των ε, πόρων. Στην έκθεση Επίπερ είχαμε ζητήσει κατανομή ένα πρόγραμμα δεν τη δέχτηκε την πρόταση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή στην περιφέρειά μου έχουν μπλοκαριστεί διάφορα προγράμματα ε, γιατί η περιφέρεια έχει ε, δαπανίσει όλους τους ε, πόρους. Η ισπανική πλευρά έχει δαπανίσει όλους τους πόρους της και επομένως έχουν μπλοκαριστεί τα προγράμματα. Αυτό είναι γελίο στο άρθρο 4 του κανονισμού εδαφικής συνεργασίας. Ε, από το άρθρο αυτό διαφαίνεται ότι η συνεργασία θα γίνει ε, ετήσια βάσει δημογραφικού κριτηρίου ε, η θεμητότητα ενός ε, έργου ε, δεν αφορά μονάχα την ε, κατανομή των κονδυλίων, κυρίως δε και πολλό δε μάλλον, όπου στο άρθρο 7 λατινικό F αναφέρεται ότι η κατανομή δεν θα γίνεται με δημογραφικά κριτήρια. Ε, επίσης ε, ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να διατηρηθεί το όριο των 150 χιλιόμετρων αλλά αναρωτιόμαστε εάν υπάρχει λόγος να διατηρηθεί αυτό το 20% maximum επένδυσης εκτός του προγράμματος. Η άλλη μου ερώτηση αφορά το ποσοστό συγχρηματοδότησης. Τι θα κάνουμε με τα, έτσι ώστε να γίνουν ελκυστικές αυτές οι διασυνοριακές επενδύσεις. Η Επιτροπή προτείνει για την εδαφική συνεργασία ένα ε, ενιαίο ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% σε όλες τις χώρες μέλη, ενώ ε, κάποιες περιοχές με ειδικούς στόχους ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας φτάνουν στο 85% η Επιτροπή μήπως μπορεί να μας δώσει αξιολόγηση του μέσου ποσοστού χρηματοδότησης που χρησιμοποιούν ε, οι ε, διαχειριστικές αρχές του προγράμματος αυτή τη στιγμή. Επίσης, συμμερίζομαι την άποψη της Ρίκα Μάνερ όσον αφορά την ε, τεχνική αρρωγή. Θεωρώ ότι θα πρέπει αναπερίπτωση και για τα μικρά προγράμματα να γίνεται επαναδιαπραγμάτευση. Η θεματική συγκέντρωση είναι καλή για να έχουμε καλά αποτελέσματα, αλλά παρόλα αυτά στο άρθρο 5 θα πρέπει να προβλέψουμε μεγαλύτερη ευελιξία συγκέντρωση 85% ε, του συνόλου σε τρία κατά προτεραιότητα προγράμματα συν την διασυνοριακή συνεργασία. Είπα και σήμερα το πρωί ότι σε αυτήν την, σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι ο μεγάλος απόν είναι η πολιτιστική δραστηριότητα. Θα πρέπει να βάλουμε περισσότερο πολιτισμό. Θα ήθελα πάντως να υπενθυμίσω όσον αφορά τον συντονισμό με το Ευρωπαϊκό Ταμείο, ε, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ε, είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει απλούστευση ε, και να ε, μπορέσουμε να έχουμε χρηματοδότηση απευθείας από το ΦΕΝΤΕΡ. Ήδη τα πράγματα είναι περίπλοκα και επομένως δεν χρειάζεται να μπλέξουμε περισσότερο. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι θα πρέπει να προσαρμόσουμε τους δείκτες στην εδαφική συνεργασία όσον αφορά τις απλουστεύσεις ε, management και ελέγχου. Κυρίως δε στο θέμα ε, της συνένωσης ε, των, επιτροπ... των αρχών διαχείρισης και επιστοποίησης ε, ε, συμφωνώ ε, εάν έχουμε όμως έναν καλό φορέα πιστοποίησης δεν θα πρέπει να τον ε, βγάλουμε ε, γιατί τότε μπορεί να υποφέρει όλο το πρόγραμμα οι εδαφικές, οι όμιλοι εδαφικής ε, συνεργασίας, ναι βεβαίως θα πρέπει να συνεχίσουν, αλλά με μεγάλη προσοχή. Επίσης θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά τις επικαλύψεις. Τέλος, δεν νομίζω ότι υπάρχει χρόνος ε, για να προετοιμαστούν σωστά τα επιχειρησιακά προγράμματα. Ενδεχομένως θα πρέπει να ξαναδούμε το χρονικό, τη χρονική προθεσμία. Τελειώνοντας να ευχαριστήσω την κυρία Μάνερ ε, για τη συνεργασία της και βεβαίω είμαι πάντα στην διάθεσή της. Ευχαριστώ πολύ. Φρανσουά Ευχαριστώ. Σχετικά με την έκθεση αυτή Πιστεύω ότι καταρχάς είναι ανάγκη να αντιληφθούμε ότι οι, οι καταστάσεις διαφέρουν κατά περίπτωση και τα προγράμματα που πρέπει να εφαρμοστούν για την διασυνοριακή συνεργασία διαφέρουν αναλόγως ε, από το εάν βρίσκεται κανείς στην πεδιάδα, στο βουνό, κοντά στη θάλασσα, στην ενδοχώρα κτλ. Ως εκ τούτου και ε, θεωρώ ότι είναι παρακινδυνευμένο να προσπαθήσουμε ε, να ακολουθήσουμε τις συλλογιστική των ε, θεματικών συγκεντρώσεων που θα ε, αποδυναμώσουν την τοπική δραστηριότητα και να κοιτάξουμε να έχουμε ε, να χρησιμοποιήσουν άξονες την διασυνοριακή συνεργασία στο πλαίσιο του ΦΕΝΤΕΡ. Αν και δεν είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουμε. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα επιτύχουμε μεγαλύτερη ευελιξία ευελιξία. Ένα άλλο θέμα που με απασχολεί και απασχολεί όλους τους νησιώτες είναι ότι η ιδέα των συνερών είναι μία χερσαία αντιμετώπιση και ε, ε, η ιδέα των 150 χιλιόμετρων ε, δεν είναι σαφές διότι ένα νησί μπορεί να είναι πολύ απομακρυσμένο από την ενδοχώρα και τουλάχιστον πρέπει να εξαιρέσουμε τα νησιά από αυτή την αρχή διότι τότε στην περίπτωσή μου η Κορσική δεν θα μπορούσε να συνεργαστεί με τις Βαλεαρίδες κάτι το οποίο θα ήταν πολύ οξύμορο σαν επίπτωση γι' αυτό και επιμένω γιατί όλες οι νησιωτικές περιοχές θα πρέπει οι ίδιες να μπορέσουν να καταρτήσουν τα προγράμματά τους διασυνοριακής συνεργασίας. Άλλωστε, το ποσό των πιστώσεων που δίδεται σε αυτήν τη διασυνοριακή συνεργασία από την Επιτροπή είναι ε, πολύ περιορισμένο. Το Κοινοβούλιο είχε καθορίσει ένα σωστό στόχο που ανταποκρινόταν στους στόχους και στα μέσα τα οποία έχουμε καταρτήσει και η αύξηση των μέσων θα αυξήσει και τις ανάγκες και αν θελήσουμε να αξιοποιήσουμε κάθε ευρώ της Ευρώπης το οποίο επενδύεται στα προγράμματα θα δούμε ότι αυτά που έχουν την καλύτερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία είναι αυτά που θα αποδώσουν περισσότερο και θα πρέπει να προσανατολιστούμε διαφορετικά από ό,τι μέχρι τώρα. Πρόκειται για μία πρόοδο, δεν το αμφισβητώ, αλλά η πρόοδος αυτή είναι ανεπαρκής μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ. Κύριε Μάρτιν, θέλετε να μιλήσετε, το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επανέρχομαι στα συγκεκριμένα θέματα που εφήγησαν. Η έκθεση είναι πολύ σαφής και η παρουσίαση ήταν πολύ σαφής. Σχετικά με την ε, ε, πολλαπλή συγχρηματοδότηση και γιατί αποκλείεται ε, στο άρθρο 88 του κανονισμού θα πρέπει να εξετάσετε τον αρμόδιο κανονισμό που δίδει μεγαλύτερη ευελιξία και άρα γι' αυτό το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι αναγκαίο να υπάρξουν αυτές οι διατάξεις διότι ήδη στον κανονισμό ε, για την ε, ε, δαφική συνεργασία προβλέπονται προτεραιότητες για τις επενδύσεις οι οποίες συνάδουν με τον με ε, το πλαίσιο, το κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Άρα χρειάζεται να υπάρχει μία πολλαπλή επένδυση. Δεν είναι ένας μηχανισμός ο νέος που χρειάζεται, άπαξ και έχει καταρτιστεί με την παραπομπή σε αυτές τις προτεραιότητες. Επανερχόμενος στο θέμα της θεματικής συγκεντρώσεως υπάρχουν, ε, χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη ευελιξία για, το, ε, ε, για τη διασυνοριακή συνεργασία από ότι για το ευρωπαϊκό περιφερειακό πλαίσιο για ε, ε, διότι οι θεματικές στόχοι διαφέρουν και δεν περιλαμβάνονται στους 11 στόχους διασυνοριακής συνεργασίας. Και σας είπα ότι με αυτή τη μεγαλύτερη ευελιξία για τις διασυνοριακές επενδύσεις το θέμα αλλάζει. Πέραν αυτού όμως αυτό το σκεπτικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να ισχύσει και για την διασυνοριακή συνεργασία να γίνουν δηλαδή σωστές επιλογές από τα προγράμματα κατά τρόπον ε, ώστε να ε, ε, εντοπίσουμε τους στόχους και να γίνονται οι σωστές επενδύσεις. Θεωρούμε λοιπόν ότι δεν πρέπει να υπάρξει αποδυνάμεση του στόχου αυτού, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ του επίπεδου συγκεντρώσεως και του ύψους της χρηματοδοτήσεως και στα πλαίσια του τωρινού μας προγράμματος για τα EOS θεωρούμε ότι ε, αντιμετωπίζουμε ε, επαρκώς τις ανάγκες και με τις τέσσερις θεματικές ενότητες δεν θέλουμε να οδηγήσουμε σε έναν αμοιβαίο αποκλεισμό, πράγμα το οποίο θα δημιουργούσε προβλήματα. Τώρα, για την κατάργηση της μεταφοράς 15% μεταξύ ε, των περιφερειών που ισχύει στο τωρινό σχέδιο. Ο λόγος για τον οποίο δεν υιοθετήσαμε αυτή τη δυνατότητα είναι ότι υπάρχει επιπρόσθετη χρηματοδότηση γενικώ και άρα ε, μπορεί να υπάρξει ε, εντός της χώρας κατανομή των πόρων και δεν υπάρχει λόγος να επέμβουμε διασυνοριακά και υπάρχει δυνατότητα να γίνουν όλες αυτές οι προσαρμογές. Τα επίπεδα τα οποία εφαρμόζονται γενικώ συνήθως είναι κάτω από το ανώτατο επίπεδο, είναι μάλλον περιορισμένα και έτσι στην γενική αυτή προσέγγιση θεωρούμε ότι υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο προστίθεται ένα νέο στοιχείο εδώ και αυτό ήταν και το σκεπτικό μας για τον τρόπο με τον οποίο καταρτίζονται τα προγράμματα είναι ότι ξεκινάμε με τις αναθέσεις ε, κατά κράτος μέλος ανάλογα του ΕΟΕΣ και μετά ε, το κάθε κράτος μπορεί να επιλέξει ποια ε, διασυνοριακά προγράμματα θα προωθήσει. Αυτό έχει σχέση με τη δομή των προγραμμάτων και οδηγεί σε διαπραγματεύσεις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών για να αποφασίσουν ποιοι τομείς των προγραμμάτων πρέπει να προωθηθούν. Έπρεπε να δούμε εάν πρέπει να υπάρχει ε, ανάθεση των προγραμμάτων, αλλά αυτό θα δημιουργούσε προβλήματα και πάλι θεωρήσαμε ότι δεν δικαιολογεί το η προσπάθεια αυτή στο, στην ισχύουσα κατάσταση. Άπαξ και τα προγράμματα όπως προβλέπονται στον κανονισμό επιτρέψουν να ληφθεί μία απόφαση και άπαξ και ληφθεί αυτή η απόφαση τότε θα πρέπει ε, να ε, ε, εξετάσουμε πού ανατίθενται τα προγράμματα πιο συγκεκριμένα για το όριο των 150 χιλιόμετρων. Υποθέτω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο συν, ε, να δούμε συχνά διότι για τα προγράμματα η ένδειξη διασύνοριακά είναι ότι αναφέρονται σε περιοχές όπου υπάρχει ε, υπάρχουν χερσαία σύνορα μεταξύ δύο περιοχών για να ε, προωθήσουμε τις παραμεθόριες περιοχές και να μπορέσουμε να προωθήσουμε τις διασυνοριακές επενδύσεις και την σχετική οικονομική ανάπτυξη. Αν έχετε θαλάσσια σύνορα τότε η κατάσταση είναι διαφορετική και οι προποθέσει είναι διαφορετικές. Γι' αυτό θεωρούμε ότι σε κάποιο σημείο δεν μπορεί πλέον να θεωρήσει ότι μπορεί κανείς να προσωμιάσει τα σύνορα, τα θαλάσσια σύνορα με τα χερσαία σύνορα. Και Γι' αυτό τώρα υπάρχει ένα όριο 150 χιλιόμετρων. Ό,τι όριο λοιπόν και να επιλεχθεί πάντοτε θα υπάρχει μία δύσκολη κατάσταση διότι θα το έχετε ξεπεράσει. Αλλά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε αποφασίσει, το διατηρούμε διότι αν δεν το χρησιμοποιήσουμε πού θα πάμε και αν δεν υπάρχει όριο θα αποδυναμώσουμε την ε, ιδέα αυτή της διεθνής εθνικής συνεργασίας η οποία προωθεί τη συνεργασία μεταξύ περιοχών που δεν είναι σε θέση να υποφεληθούν από τη διασυνοριακή συνεργασία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ε, ποσοστό συγχρηματοδότησης. Η προσέγγιση ήταν ακριβώς να απλουστεύσουμε, να έχουμε ένα μόνο συντελεστή συγχρηματοδότησης. Διατηρείται σε υψηλό επίπεδο Σίγουρα θα υπάρχει δυνατότητα να αναλύσουμε τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας και να βρούμε στοιχεία για το μέσο όρο συγχρηματοδότησης ε, και τι γίνεται εκεί, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό είναι συνιστά πλούστευση. Δεν πάει κατά περίπτωση η εξέταση ποια θα ε, πρέπει να είναι τα επίπεδα συγχρηματοδότησης ανάλογα με το έργο. Και νομίζω ότι αυτό είναι καλό. Γιατί δεν αποθαρρύνει τις επενδύσεις που θα μπορούσε σε αντίθετη περίπτωση. Σε ό,τι αφορά τη διαχειριστική τη, ε, ε, αρχή που δίνει την αδειοδότηση ή πιστοποίηση. Κάποια στιγμή θα πρέπει να επιβάλλουμε μια απλοποίηση, γιατί υπάρχουν κάποιοι τομείς που μπορεί κάτι να φαίνεται γενικά απλοποίηση, αλλά ένα κράτος μέλος δεν το θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει την πρόθεση να υλοποιήσει αυτά που ε, πρότεινε και που έχει φροντίσει να προωθηθούν για τους δικαιούχους. Ένα από τα στοιχεία αυτά είναι το θέμα της απλοποίησης. Πραγματικά θέλουμε να το διατηρήσουμε. Θεωρούμε ότι στα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας δεν θα πρέπει να υπάρχει χωριστή αρχή ε, πιστοποίησης. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία. Εδώ δεν τη βλέπουμε σχέση με άλλα προγράμματα γιατί ακριβώς είναι πολύ διαφορετικές οι ρυθμίσεις για τη διαχείριση, τον έλεγχο, για τις ε, ροές και τις εκταμιεύσεις. Σε άλλες περιπτώσεις μπορούν να είναι χωριστές αυτές οι δύο αρχές, ενώ στη συγκεκριμένη ε, μπορεί να είναι η ίδια. Διαχείριση και επιστοποίηση στον ίδιο φορέα. Αυτά νομίζω ήταν τα συγκεκριμένα ερωτήματα που μου είχαν απευθύνει. Ο κύριος Χρυσόγελος, παρακαλώ, σύντομα σχόλιο και μετά προχωρούμε. Yes, θα ήθελα να επανέλθω στο 13 για το Ταμείο Συνοχής. Όχι τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι μίλησαν. Πολύ χρήσιμα ήταν τα σχόλιά σας και θα με βοηθήσουν πολύ ε, στη δουλειά μου, ιδιαίτερα και ε, τα θέματα των λεπτομεριών θα τα συζητήσουμε με τους και ε, και θα τα διαπραγματευτούμε την ησυχία μας και σίγουρα θα βρούμε κάποια λύση. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια. Αυτός ο χιλιομετρικός περιορισμός. Άκουσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό μαζί τους. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο όριο, 50 χιλιόμετρα. Μου φαίνεται αρκετά δικαιολογημένο αυτό. Κάπου δεν θα πρέπει να βάλουμε ένα όριο μέχρι πού θα φτάνει η εδαφική συνεργασία. Συμφωνώ με την Κομισιόν. Αυτό βεβαίω προκαλεί κάποια προβλήματα, όπω είπε ο κύριο Αλφόνση, σε περίπτωση νησιών. Ε, δεν θα το κοιτάξουμε αυτό, θα το σκεφτούμε. Ε, κάποια λύση θα βρούμε και για τα νησιά. Με κάποια τροπολογία ή τροποποίηση, εν πάση περιπτώσει, έτσι ώστε να καλύπτονται ειδικέ περιπτώσει και να εντάσσονται για τις αναθέσεις αναέργο. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία όλοι ακούσαμε, θα πρέπει να το συζητήσουμε διμερώς, νομίζω αξίζει τον κόπο. Πάντως, όταν ε, ανατίθεται στα κράτη-μέλη, τα κράτη αποφασίζουν με βάση κριτήρια ε, πληθυσμιακά δεν θα πρέπει να είναι μόνο κατά πόσο είναι πυκνοκατοικημένη ή αεροκατοικημένη μια περιφέρεια. Αυτά προς το παρόν. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ. Μπορούμε να επανέλθουμε στο 13 που είχαμε διακόψει πριν το μεσημέρι το Ταμείο Συνοχής και ε, ο Νίκος Χρυσόγελος νομίζω θέλει το λόγο για να μιλήσει για το 13. Και μετά, Βίκτορ, αν θέλεις να ολοκληρώσεις. Όχι, θα ήθελα μόνο ο κύριος Μποστινάρου να προτείνω κυρία Πρόεδρε και σε όλους τους αξιότιμους συναδέλφους, επειδή είμαστε πάρα πολύ λίγοι αυτή τη στιγμή στην αίθουσα, ή δυνατόν, ε, αν είναι απαραίτητο, είμαι στη διάθεσή σας να σας ακούσω και να απαντήσω στις ερωτήσεις. Αλλιώς, να συνεχίσουμε ε, σε άλλη ευκαιρία, άλλη στιγμή, αν συμφωνήσετε, να μπει στην ημερήσια διάταξη το θέμα. Αλλά να ακούσω τις ερωτήσεις ή τα σχόλια των εκλεκτών συναδέλφων μας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, μερικές παρατηρήσεις εκ μέρους ομάδας των ε, Πρασίνων. Ε, με δεδομένο ότι η πολιτική συνοχή δεν αποβλέπει μόνο στην πρόθεση της οικονομικής ε, μεγένθησης και της κοινή αγοράς, αλλά κατά βάση στην κοινωνική συνοχή και στην περιβαλλοντική συνοχή, νομίζω ότι το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να δώσει μεγάλη έμφαση στη συνοχή μεταξύ των επιμέρων στόχων, ε, αφενός μεταξύ των διαφόρων θεματικών προτεραιοτήτων, ώστε να μην αντιφάσκει μία με την άλλη, δηλαδή να υπάρχει μια και οριζόντια συνεργασία μεταξύ των τομέων των προτεραιοτήτων θεματικών, αλλά και από την άλλη μεριά να διευκολύνει την προώθηση υποδομών που αντιστοιχούν και είναι κατάλληλε για την κάθε περιφέρεια. Δηλαδή, κάθε περιφέρεια έχει ιδιαιτερότητε και γι' αυτό οι υποδομέ, θα αφορούν την ενέργεια, είτε το περιβάλλον, είτε τι μεταφορέ, πρέπει να είναι ε, προσαρμοσμένε στι δυνατότητε και στι προτεραιότητε αυτών των περιοχών. Αλλιώ είναι πιθανό ότι έχουμε σπατάλη πόρων και αναποτελεσματικότητα. Ε, Ήθελα να τονίσω επίσης ότι οι πολιτικές συνοχής ε, αφορούν βέβαια συνοχή μεταξύ περιφερειών της Ευρώπης, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα και μέσα σε αναπτυγμένες περιοχές, περιφέρειες, υπάρχουν πολλές ανισότητες και υπάρχουν περιοχές hot spots που ε, αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα. Άρα Προφανώς πρέπει να υπάρχει συνοχή μεταξύ των διαφόρων περιφερειών της Ευρώπης, αλλά να δώσουμε έμφαση και στο εσωτερικό κάθε περιφέρειας τώρα, νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή, έτσι ώστε να καλύψουμε τις εσωτερικές διαφορές και ανισότητες. Και εκεί να επικεντρώσουμε κατάλληλα τους πόρους. Ε, ήθελα να τονίσω επίσης και μετά την εισήγηση της μελέτης ε, που ακούσαμε πριν λίγο τα δεδομένα της οικονομικής κρίσης αλλάζουν και το στάτους, το καθεστώς των περιφερειών. Ήδη ακούστηκε ότι τρεις από τις ελληνικές περιφέρειες, με βάση τα στοιχεία του 2009, ε, πέφτουν στην κατηγορία των ανδιάμεσων ε, περιφερειών, υπομετάβαση. Ε, είμαι σίγουρος ότι αν δούμε τα στοιχεία του 10 και του 11 και του 12, αυτό θα αλλάξει δραματικά γιατί έχουμε αύξηση της ανεργίας, έχουμε αύξηση της ε, φτώχειας και έχουμε και μείωση δραστική του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε διάφορες περιοχές. Επομένως, δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε τη στρατηγική 2014-2020 με στοιχεία πρώτης κρίσης. Θα πρέπει να το πάρουμε σοβαρά υπόψη και να προσαρμόσουμε τα κριτήρια για, με βάση τα νέα δεδομένα που έχουμε για αυτές τις περιοχές. Ε, ήθελα επίσης να τονίσω ότι δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση και πολύ σωστά στην, ε, στο ρόλο μπορούν να παίξουν οι πόλεις και στα θέματα συνοχής και στα θέματα προστασίας του κλίματος και προστασίας του περιβάλλοντος. Είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί μεγάλο ποσό του πληθυσμού ζει στις πόλεις. Και εκεί υπάρχει και τεράστιο δυναμικό να βελτιώσουμε τις περιβαλλοντικές μας επιδόσεις. Από την άλλη μεριά όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι προβλήματα συνοχής αντιμετωπίζουν ορεινές περιοχές και ιδιαίτερα νησιά. Ακόμα και αν αυτά φαίνεται ότι έχουν υψηλό ακαθάριστο εθνικό προϊόν, αυτέ οι περιοχέ αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα λόγω των ιδιαιτεροτήτων του στα θέματα συνοχή. Ε, έτσι λοιπόν και σε γενικέ γραμμέ αλλά και σε ειδικά εργαλεία θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τι περιοχέ αυτέ. Για παράδειγμα, το Connecting Europe Facility θα πρέπει να λάβει υπόψη και τη σύνδεση όχι μόνο μεταξύ περιφερειών ή διασυνοριακέ συνδέσει, αλλά θα πρέπει να πάρει υπόψη και τη σύνδεση μεταξύ νησιών και βέβαια και ορεινών περιοχών γιατί υπάρχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα σύνδεση μεταξύ νησιών και θα έλεγα ότι δεν αφορά μόνο τους κατοίκους, μόνιμους κατοίκους των νησιών, αφορά όμως και Ευρωπαίους πολίτες από άλλες περιοχές, από άλλες περιφέρειες που επισκέπτονται αυτά τα νησιά και όχι μόνο το καλοκαίρι. Θα θέλουν να επισκεφθούν αυτά τα νησιά. Άρα οι πολιτικές μας, όταν μιλάμε για, την, ε, για τις μεταφορές, πρέπει αφενός να στοχεύουν στη βιώσιμη κινητικότητα, όχι μόνο σε βαριές υποδομές αυτοκινητοδρόμους, αλλά και βιώσιμη κινητικότητα μέσα στις πόλεις και παράλληλα ε, συνδέσεις κατάλληλες, ιδιαίτερα με έξυπνα και πράσινα μέσα μεταφοράς, δηλαδή έξυπνα σκάφη, μεταξύ νησιωτικών και παράκτων περιοχών. Και εκεί υπάρχει ένα τεράστιο πεδίο συνοχής με τις πολιτικές για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις που αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως για παράδειγμα για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του αζότου, διοξιδίου του θείου ή τις τιμίες των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Άρα λοιπόν εκεί θέλουμε μεγαλύτερη έμφαση σε αυτές τις πολιτικές συνοχής. Είμαστε σίγουρα υπέρ πολιτικών που αντιμετωπίζουν τα δημοσιονομικά προβλήματα στις χώρες που έχουν σοβαρά προβλήματα. Δεν πρέπει όμως αυτές οι πολιτικές να δημιουργήσουν δυσκολίες στο να προσαρμοστούν οι περιφέρειες και να βελτιώσουν τις ε, επιδόσεις τους στη συνοχή. Δηλαδή να μην έχουμε πολιτικέ τιμωρία αυτών των περιοχών, αλλά διευκόλυνση μέσα από εκπαίδευση, μέσα από κατάλληλη υποστήριξη, ώστε να πετύχουν πραγματικά τη συνοχή και όχι να τιμωρηθούν γιατί πιθανά υπάρχουν δημοσιονομικά προβλήματα. Ένα σημαντικό επίση θέμα είναι το θέμα των εταιρικών σχέσεων, το partnership contracts. Ε, θα θέλαμε να δούμε συναπόφαση, συναρμοδιότητα μεταξύ κεντρικών κρατών και περιφερειών και τοπικών αυτοδιοικήσεων και βέβαια σε αυτό το διάλογο να παίρνουν μέρος και οι κοινωνικοί εταίροι, οι stakeholders σε τοπικό επίπεδο, γιατί έτσι μπορούμε να διαμορφώσουμε πραγματικά προτεραιότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ενδυναμώσουμε αυτή την έννοια της εταιρική σχέσης, ίσως και με θεσμικό τρόπο, μέσα από μια λογική συναπόφαση κεντρικού κράτους, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περιφερειακών αρχών και, και βέβαια και περιφερειακών συμβουλίων, για να υπάρχουν πραγματικά μεγαλύτερη συνοχή. Ε, και τέλος θα ήθελα να πω ότι για το ε, Connecting Europe Facility ε, είμαστε υπέρ εάν επικεντρώσει, όπως είπα πριν, και σε συνδέσεις μεταξύ νησιών, αλλά κυρίως σε συνδέσεις με σιδηροδρομικές γραμμές μεταξύ των περιοχών. Να μην συνεχίσουμε να επενδύουμε υπερβολικά πολύ σε αυτοκινητοδρόμους που δημιουργούν και άλλα προβλήματα, όχι μόνο περιβαλλοντικά. και θα ήθελα να προτείνω και, και τέλος και μια ε, ρύθμιση μοιάζει λίγο βέβαια ε, υπερβολική σε κάποιους, αλλά νομίζω ότι είναι απαραίτητη σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα που έχουν σοβαρά προβλήματα χωροταξικού σχεδιασμού. Να συνδέσουμε τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής και με την υποχρέωση των περιφερειών και των κρατών να ολοκληρώσουν το χωροταξικό σχεδιασμό και τις χρήσεις γης σε αυτές τις ε, περιοχές γιατί πολλές φορές η απουσία χωροταξικών σχεδίων δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα πραγματικά περιβαλλοντικής συνοχής και έχουμε αντίφαση μεταξύ πολιτικών συνοχής που δημιουργούν υποδομές και έργων τα οποία γίνονται, τα οποία καταστρέφουν το περιβάλλον. Άρα πρέπει να ενισχύσουμε αυτή την έννοια της συνοχής και σε αυτό το επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. You mentioned so many issues ε, ε, Βίκτορ, θέλεις να απαντήσεις, ανέφερες ε, τόσα πράγματα. Λοιπόν, να απαντήσω. Ειλικρινά πιστεύω ότι το Ταμείο Συνοχής δεν μπορεί να είναι το σακούλι του Άγιου Βασίλη. Δεύτερον, υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Ε, ε Βεβαίω, καλωσορίζω την ιδέα ότι χωρίς ε, σημαντικό προϋπολογισμό ε, για την πολιτική συνοχή οι ιδέες μας και τα σχέδιά μας και οι εκθέσεις μας όταν και εφόσον εγκριθούν θα παραμείνουν στοιχεία θεωρητικού διαλόγου άνευ πραγματοποιήσεως και υλοποίησεως. Άρα ναι, πρέπει να υπάρχει σημαντικός προϋπολογισμός. Τρίτον, αμφιβάλλω σοβαρά σχετικά με το κάπινγκ, σχετικά με την μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Ε, δεν δέχομαι την ιδέα αυτή. Επίσης με απασχολεί πολύ αυτό το αποθεματικό απόδοσης ε, και νομίζω ότι προς τα εκεί συγκλίνουν και οι εμπειρογνώμονες που ακούσαμε το απόγευμα ε, στοιχεία, πληροφορίες, στατιστικά συμφωνώ και εγώ ότι με την κρίση ε, θα μεγαλώσει το, η διάσταση μεταξύ πτωχών και πλουσίων περιφερειών. Οι φτωχές θα γίνουν φτωχότερες και ενδεχομένως οι πλούσιες πλουσιότερες. Ειλικρινά και για να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια από τα ζητήματα τα οποία αναφέρθηκαν, να πω ότι Συμφωνώ απολύτως με το άνοιγμα της ε, δυνατότητας εξοικονόμησης ενέργειας ε, για τα νοικοκυριά ε, σε σχέση και με την ενεργειακή αποδοτικότητα, απόδοση καθώς επίσης και με την κλιματική αλλαγή και ε, ώστε να αντιμετωπίσουμε και την εκπομπή ρήπων και αερίων του θερμοκηπίου. Επίσης, ε, συμφωνώ να βάλουμε στην ε, συζήτησή μας τα, τις εγκαταστάσεις ενέργειας καθώς επίσης και όλα αυτά τα προγράμματα περιφερειακής διανομής ενέργειας. Τώρα το μέσο Connecting Europe ε, νομίζω πως είναι η απάντηση στα προβλήματα τα οποία ε, σχετίζονται με την διασυνοριακή διασύνδεση και όχι μόνο. Πρέπει να αποφασίσουμε ε, επί σαφών και αξιοπρεπών κανόνων που θα μας βοηθήσουν έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα και ειδικά προβλήματα κάποιων συγκεκριμένων χωρών που εκφράστηκαν ήδη. Τέλος, Συμφωνώ απολύτως η κλιματική και η, ε, κλιματική αλλαγή να ενταχθούν στους κανόνες εταιρικής σχέσης, σχέσης μας. Ε, τα, οι παράμετροι αυτοί όχι μόνο να ληφθούν υπόψη αλλά ε, να ε, απαντηθούν σωστά από, τις, από τους εμπλεκόμενους φορείς ούτως ώστε αυτοί να γίνουν επιλέξιμοι. Γι' αυτό λοιπόν θα ζητήσω και από τον Επίτροπο Ποτόσνικ όσο γίνεται πιο γρήγορα να μας υποβάλει την ε, το τροποποιημένο ε, κείμενο σχετικά ε, με τις μελέτες επιπτώσεων. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να κρατήσουμε και κάποια ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και την ανάγκη να παραμείνουν ανθρώπινες οι πόλες μας ανάμεσα στην ανάγκη θέρμανσης αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακος και λοιπόν εκπομπών, αλλά όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, λοιπόν όλα αυτά ήθελα να πω, ε, υπάρχουν βέβαια και κάποια όρια, εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ, θα κάνω όλες τις προτάσεις και με τη δικιά σας αρρωγή και τις δικές σας συνεισφορές βεβαίως θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα εδώ να τελειώσουμε τη συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ. Αναβάλαμε το θέμα της στέγασης για την επόμενη συνεδρίαση ραντεβού στις 26 Απριλίου. Ε, είναι δύο μισές μέρες, είναι μικρότερη συνεδρίαση από αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστώ, λήξη συνεδρίαση. Χαίρετε.